Sí. Le ruego que vayan tomando... Παρακαλώ καθίστε. Καθίστε για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Bueno, pues, eh, buenas tardes. Καλησπέρα σας λοιπόν. Καλησπέρα. Σήμερα έχω τη χαρά να καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο στόχος που μας απασχολεί σήμερα, που είναι η συζήτηση των θέσεων των διαφόρων κοινοβουλίων για την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, είναι αρκετά σημαντικός, ώστε να μαζευόμαστε εδώ όλοι για πρώτη φορά για να συζητήσουμε θέματα αλληλείας θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε σήμερα 38 μέλη από 23 κοινοβούλια, τα οποία εκπροσωπούν 19 κράτη-μέλη και φυσικά θα ήθελα να καλωσορίσω και την Επίτροπο Αρμόδια για θέματα ναυτιλίας και αλληλείας, την κυρία Οδαμανάκη, και να την ευχαριστήσω διότι κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα για να μας πει και το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο τη διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε και ελπίζω να μην είναι αρκετά ε, προβληματική ώστε να μπορέσετε όλοι να ε, λάβετε το λόγο. Στον πρώτο γύρο συζητήσεων, επαναλαμβάνω στον πρώτο γύρο, μετά από την κυρία Δεμιανά και την κυρία Πατράου που θα μιλήσουν εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, θα καλέσω έναν εκπρόσωπο από κάθε κοινοβούλιο Δηλαδή, στην περίπτωση που έχουμε δύο διαφορετικά κοινοβούλια ε, σε μία χώρα, θα έχουμε έναν εκπρόσωπο από κάθε κοινοβούλιο και θα τους δώσουμε το λόγο για τέσσερα λεπτά, προκειμένου να παρουσιάσουν τη θέση του κάθε κοινοβουλίου. Ένας λοιπόν αναβουλή σε περίπτωση που έχουμε εκπροσώπους από δύο διαφορετικές βουλές ε, μίας χώρας θα έχουμε έναν για κάθε βουλή. Ε, σας έχει διανεμηθεί το έντυπο που έχω εδώ μπροστά μου και θα ήθελα να σημειώσετε το όνομα του εκπροσώπου που θα μιλήσει για κάθε κοινοβούλιο. Τώρα θα περάσουν οι κλητήρε να το ε, πάρουν και σας παρακαλώ να σημειώσετε τα ονόματα αυτών που θα μιλήσουν. Εάν κάποιος εκπρόσωπος από κάποιο κράτος μέλος δεν θέλει να λάβει το λόγο, δεν υποχρεούται φυσικά να το κάνει. Γι' αυτό ακριβώς δίδεται το έντυπο για να σημειώσετε ποιος θέλει να μιλήσει και εκ μέρου ποιου κοινοβουλίου. Και στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή θα έχουμε ακούσει τους εκπροσώπους από κάθε κοινοβούλιο θα ξεκινήσει μια συζήτηση στην οποία θα δοθεί δυνατότητα στους υπολείπους εκπροσώπους να παρέμβουν καθώς επίσης και στους ευρωβουλευτές. Για να ε, γίνει αυτός ο δεύτερος γύρος ομιλίας θα σας δοθεί δεύτερο έντυπο. Επομένως, στον πρώτο γύρο σας παρακαλώ σημειώστε στο έντυπο μόνο τους εκπροσώπους από κάθε κοινοβούλιο και θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος, θα σας δοθεί δεύτερο έντυπο και σας παρακαλώ να σημειώσετε εκεί ποιο, ε, είτε από το Ευρωκοινοβούλιο είτε από τα υπόλοιπα κοινοβούλια θέλει να λάβει το λόγο. Να σας πω επίση ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται απευθείας ε, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πλέον χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να δώσω το λόγο στην Επίτροπο κυρία Δαμανάκη η οποία θα σας μιλήσει για περίπου 10 λεπτά. 10 ε, λεπτά το πολύ θα ήθελα να σας ζητήσω. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Δαμανάκη, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. κυρίες και κύριοι βουλευτές των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίων. Δεν συναντώ συχνά από κοινού εθνικούς και ευρωβουλευτές. Και αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα. Πάνω απ' όλα διότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας ε, φέρνει στο δρόμο μιας νέας και ενισχυμένης συνεργασίας. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ένα πλήρη ρόλο, πληρέστερο ρόλο για πολλούς τομείς από ό,τι πριν. Οι εθνικές βουλές επίσης έχουν αναβαθμισμένο ρόλο. Σήμερα θα ήθελα να σας δώσω μια ιδέα του πού βρισκόμαστε ως προς τη συζήτηση για την αναθεώρηση της κοινή αλλιευτικής παλιτικής και των θεμάτων που θέτει. των θεμάτων που τίθενται και κατά τη διαβούλευση και κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις μας με τους ενδιαφερόμενους μεταξύ των οποίων και στο περασμένο άτυπο συνέδριο των Υπουργών Αλληλείας στο Βίγκο της Ισπανίας. Ας αρχίσω με τα περιφερειακά. Η ιδέα περιφερειακών οργανώσεων ή υπηρεσιών όπου να, κατανέμ, όπου να κατανέμεται η διοργάνωση είναι, δεν είναι καινούργια, αλλά το σαφές είναι ότι πρέπει να έχουν αποτελέσματα και όχι να δημιουργηθούν νέες δομές μόνο και μόνο για να υπάρχουν στα χαρτιά. Τα σχέδια αυτά περιφερειοποίησης θα οργανωθούν με βάση τα κράτη-μέλη και θα περιλαμβάνουν εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, της βιομηχανίας κλπ ώστε να αντικατοπτρίζουν σαφώς την τοπική πραγματικότητα και γι' αυτό υπάρχουν τα περιφερειακά συμβουλευτικά σώματα έτσι ώστε ο διάλογος και η συζήτηση να φτάσει μέχρι τις περιφέρειες, πράγμα που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε και την ποιότητα της διαχείρισής μας και την αξιοπιστία μας. Η περιφερειοποίηση λοιπόν σημαίνει ότι φτάνουμε μέχρι τον Αλιέα και την Αλιέα. Πρέπει να βρούμε τρόπους λοιπόν η βιομηχανία να συμμετάσχει και αυτή και ε, βρίσκομαι εδώ μεταξύ άλλων για να ακούσω και τις απόψεις σας για αυτό το θέμα. Άλλο θέμα τώρα. Μερικοί από εσά μπορεί να αναρωτηθείτε τι σημαίνει για μας η περιφερειοποίηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ θα ήθελα να σας πω σαφώς ότι βεβαίως οι κυριότερες κατευθύνσεις της πολιτικής αυτής θα συναποφασιστούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραδείγματος χάρη. Τα μακροπρόθεσμα προγράμματα και η καθορισμός των στόχων τους θα συναποφασίζονται με, το, με τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μεγέθη των οφθαλμών των δικτύων επίσης. Οι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι τα προσωρινά κλεισίματα περιφερειών, αλλιευτικών περιφερειών θα συναποφασίζονται. Όλα αυτά είναι παραδείγματα, όχι εξαντλητικά. Και τώρα η διάσταση της αγοράς της κοινής αλληλευτικής πολιτικής εδώ θέλουμε μεγαλύτερη ευθύνη των οργανώσεων των παραγωγών. Πρέπει να μπορέσουν να συνδεθούν καλύτερα με τις ανάγκες της αλλιευτικής αγοράς, στην οποία προμηθεύουν υψηλής ποιότητος προϊόντα. Βεβαίως, πρέπει να δούμε και ποια θα μπορούσε να είναι η καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των δημοσιονομικών. Και άρα να απαλλαχθούμε από τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις καταστροφές αλλιευμάτων. Ιδιαίτερα διότι εφόσον τα αποθέματα μειώνονται δραστικά δεν δικαιώνεται πια η καταστροφή αλλιευμάτων. Να δίνουμε χρήματα δηλαδή για την καταστροφή αλλιευμάτων. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Αντίθετα πρέπει να έχουμε μια, έναν απλό μηχανισμό αποθήκευσης που να χορηγεί καλύτερες τιμές στον αλιέα. Η βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι τα ψάρια δεν θα μπορούν να πολλούνται. αν δεν πολλούνται θα μένουν στη θάλασσα. Θα συμφωνείτε φαντάζομαι ότι πρέπει τα ίδια υψηλά πρότυπα να εφαρμόζουμε με εκείνα που ζητούμε από τους ανταγωνιστές μας και τους συμμάχους μας. Θα υπάρχει λοιπόν μια ρήτρα που θα αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά που θα είναι αναπόσπαστο τμήμα της κάλπα. Πρέπει επίσης να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Μάλλον ως τμήμα μιας τριμερούς συμφωνίας. Άλλο θέμα τώρα. Τα ITRs, Individually Tradable Rights. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο για να αποζημιωθούν ορισμένοι από τις ζημίες που υφίστανται. Και εφόσον τα αποθέματα είναι κοινό αγαθό, πρέπει να καθοριστούν τα δικαιώματα των χρηστών για περίοδο 10-15 ετών, μετά την οποία τα δικαιώματα να μπορούν να επεκτείνονται αν ο χρήστης αποδείξει ότι έχει κάνει υπεύθυνη χρήση. Αλλιώς να αποσύρονται. Τα ITR επίσης θα παίζουν και έναν δεύτερο ρόλο, δηλαδή θα μειώνουν την υπεραλίευση. Γιατί μέχρι τώρα προσπαθούσαμε να καταστρέψουμε τα αποθέματα και αυτό μας έχει απογοητεύσει διότι δεν έφερε αποτέλεσμα και παρά το ότι είναι πολύ υψηλού κόστους από την άλλη το σύστημα των ITR σε εθνικό επίπεδο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 Now, if ITR systems managed at a national level, if they are can bring down... Τώρα λέγω, αν το σύστημα των ITR έχει φέρει τόσο θετικά αποτελέσματα... Δεν... No more decommissioning of vessels with taxpayers money. Θα πρέπει να μην παραγγέλλονται πλέον, να πληρώνονται τα πλοία με τα χρήματα των φορολογούμενων βρισκόμαστε εν μέσω μιας μείζωνος οικονομικής ε, κρίσης και πραγματικά δεν βλέπω κανέναν εθνικό, εθνικό υπουργό οικονομικών, οικονομίας ο οποίος να είναι πρόθυμος να συνενέσει στη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων απόσυρσης των παλαιών πλοίων αντλώντας πόρους από τον εθνικό προϋπολογισμό για τον των, ε, του στόλου. Ε, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Το συζήτησα. Ε, και με τον τρόπο αυτό αυτή είναι θερατική καταδίκη πολλών ε, αλλιέων. Γιατί οι αλλοίς προτιμούν αυτή τη δυνατότητα ως εναλλακτική δυνατότητα αν δεν υπάρχουν άλλες ε, λύσεις. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά μια δυνατότητα μεταφοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό δεν προτίθεμαι να προτείνω τα δικαιώματα αυτά, τα ITR, να γίνονται αντικείμενο εμπορίας μεταξύ αλλιέων από διάφορε χώρες ε, μέλη. Το σύστημα των ITR, αυτών των ατομικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να παραμείνει σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή ε, και, να μην αποκτήσει διασυνοριακό χαρακτήρα. Τώρα, όσον αφορά την, της μικρής, την μικρή κλίμακος αλίας, αυτή θα πρέπει να μείνει έξω από ένα τέτοιο είδους σύστημα και θα πρέπει ε, να τοποθετείται μόνο σε μια εκούσια βάση ε, γιατί είναι ξεκάθαρο τα δικαιώματα των αλλίων μικρής κλίμακας θα πρέπει να παραμείνουν στην παρούσα διευθέτηση και να μην ισχύουν για μεγαλύτερα σκάφη και επίσης δεν θα, θα πρέπει να σευσίσουμε την προσοχή έναντι του κινδύνου της ε, υπερσυγκέντρωσης αυτών των δικαιωμάτων. Εκεί που πρόκειται για μικρά αλληλευτικά σκάφη θα πρέπει να προβλέψουμε ένα σύστημα το οποίο να, είναι πιο, να προσθέσει πιο πολλά πλεονεκτήματα γιατί αυτοί οι αλληλείς με τα μικρά σκάφη έχουν ήδη, βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική ε, θέση. Ε, από την άλλη, η δουλειά τους είναι πολύ πιο εντατική σε σχέση με τα μεγάλα ελευτικά σκάφη και δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό η ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων είναι απολύτως λογική και γνωρίζω ότι και εσείς ε, δίνετε μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο. Αλλά θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι πολλές χώρες μέλη, πολλές κυβερνήσεις εννοώ με αυτό, δεν συμφωνούν μαζί μας και δεν ε, επιθυμούν να έχουν μια ειδική προσέγγιση που να ισχύει για τα μικρά αλευτικά σκάφη. Πριν καταλήξω θα ήθελα απλώ να πω μερικά λόγια για τις υδατοκαλλιέργειες. Είναι προφανές ότι η υδατοκαλλιέργεια είναι αλληλένδετη με την κοινή ελευτική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα εντάξουμε αυτό το σημαντικό τομέα σε, αυτό, αυτή τη διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΑΛΠ. Και πραγματικά εξέτασα όλα τα σημεία που τίθενται στις εκθέσεις του Κοινοβουλίου. Και η συζήτηση αυτή μαζί σας, τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα για να ακούσω τις δικές σας απόψεις άμεσα σε σχέση με τις ε, υδατοκαλλιέργειες. Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν εδώ. Ως ε, άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι είστε σε, στην καλύτερη θέση για να εκφράσετε τις απόψεις των ψηφοφόρων σας. Και οι πολύ γόνιμες ε, συζητήσεις θα δώσουν τη βάση για τη μελλοντική συνεργασία. Δεν συμφωνούμε σε όλες τις απόψεις, αλλά συμμεριζόμαστε την επιθυμία για μια οικονομικά εύρωστη κοινή αλληλευτική πολιτική. Και είναι ακριβώς αυτό ο τομέας της Ελίας που είναι τόσο σημαντικός για τις παράκτηε περιοχές. Γιατί ε, συντηρεί περιοχές και περιφέρειες εκεί όπου μειώνονται οι θέσει εργασία στους άλλους κλάδους. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Eh, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστώ διότι θέσατε τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Πατράο Νέβες, στην οποία θα ήθελα να ζητήσω να τηρήσει τα όρια των 10 λεπτών, θα λάβει το λόγο για να σας πει ποιες είναι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι τούδε για το πράσινο Βίβλο. Κύριε Πατράου. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Αλίας, κυρία Επίτροπε, είναι χαρά να σας έχουμε εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές και να αποτανθώ και στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, στους οποίους θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την παρουσία τους εδώ. Η συνεδρίαση αυτή με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλέων, ε, η οποία είναι και η πρώτη μετά από την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και θα ήθελα να καλωσορίσω και του ε, εκπροσώπου από τα λοιπά θεσμικά όργανα και φυσικά και όλου του υπόλοιπου παρευρισκόμενου. Θεωρώ ότι ήγηκε η ώρα να εντατικοποιήσουμε τις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Πρόκειται για μια καλή ευκαιρία, διότι μετά από την έγκριση στην Ολομέλεια της έκθεσης για την πράσινη βίβλο που σχετίζεται με την ε, μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής επιτροπής, έχουμε πλέον ε, λάβει μια κάποια απόσταση και μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση πιο ήρεμη και πιο λογική για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε στο μέλλον. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία είναι πολύ συνεκτική διότι εδώ έχουμε εκπροσώπους ε, νομοθέτες ε, σε διάφορα επίπεδα που ενδιαφέρονται για αυτή τη ε, μεταρρύθμιση. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική είναι σαφέστατη και εκφράζεται και στη σχετική έκθεση η οποία έτυχε ευρεία συνένεση. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί και μια πολύ στεναρή δέσμευση για να αναλάβουμε δράση. Και προσφάτω, η έκθεση ενισχύθηκε με την έναρξη ισχύω φυσικά τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η οποία δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξουσία συναπόφαση στα θέματα αυτά μαζί με το Συμβούλιο. Επομένω, ο ρόλο του Κοινοβουλίου δεν είναι πλέον συμβουλευτικό, είναι ρόλο ε, πιο ουσιαστικό και σε επίπεδο διαπραγματευση. Οι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίστηκαν στην ευρεία συνένεση και μας οδήγησαν σε ένα διευρυμένο πλαίσιο ισορροπίας επί τη βάση και της ε, ε, εικόνας που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πλέον ξεκινά μια νέα φάση στην οποία λαμβάνουμε υπόψη και τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή προκειμένου να αναγνωριστούν με κατάλληλο τρόπο οι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Οι θέσει αυτέ ε, είναι γνωστέ ε, πλέον. Ε, μας ενδιαφέρουν ε, κάποιες στοιχειώδες άξονες και φυσικά το βλέπουμε και στους διάφορους τίτλους των κεφαλαίων της έκθεσης μια προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στα οικοσυστήματα, στα έσοδα των αλλιέων, την ε, ε, ρύθμιση των ε, αλλιευτικών επαγγελμάτων, το να γίνονται επενδύσεις και στην κατάρτιση των αλλιέων, να υπάρχει υπεύθυνο έλεγχος με διάφορα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τις ανάγκες της αλλίας και διαχείριση των στόλων κοινοτικό επίπεδο πρέπει λοιπόν να λάβουμε κατάλληλη μέρημνα ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των αλλιευτικών αποθυμάτων και στόλου, ε, υδατοκαλλιέργεια, μεταποιημένα προϊόντα. Αναγνωρίζετε το γεγονός ότι η χθεοκαλλιέργεια μπορεί να μας ε, οδηγήσει σε ποιοτικά προϊόντα τα οποία είναι συμπληρωματικά της αλληλείας ε, και επίσης ε, η κατάλληλη ε, μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων και ρόλος λοιπόν των κοινών οργανώσεων αγοράς, ε, σχέσεις ε, ε, με τρίτες χώρες, αλληλευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες οι οποίες θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και φυσικά κοινή θαλάσσια πολιτική ολοκληρωμένη στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού αλληλευτικού χώρου ο οποίος θα φροντίζει τα συμφέροντα της αλίας. Από αυτά τα οκτώ μεγάλα θέματα θα ήθελα να σταθώ κυρίως σε τρία τα οποία θεωρώ ότι αποτελούν προτεραιότητα δεδομένης της παρούσας κατάστασης. Καταρχάς αναφέρομαι στην περιφερειοποίηση ή στην αποκέντρωση. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή είναι μια πρόταση την οποία έχουμε στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόταση η οποία ε, έτυχε ομόφωνης αποδοχής από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάποιες από τις παρεμβάσεις της Επιτρόπου αλλά και σε παρεμβάσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημάνθηκαν οι δυσκολίες από νομικής πλευράς που σχετίζονται με την ενεργοποίηση αυτής της περιφερειοποίησης και την υλοποίησή της και στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Ορισμένες φορές ακούσαμε ε, και για κάτι αδύνατο το οποίο ε, δεν μπορεί να μας βοηθήσει να φτάσουμε στην εναρμόνιση. Όμως έχουμε δεσμευτεί όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και μόλις το ακούσαμε και από την ε, Επίτροπο. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάποιες σκέψεις επί του θέματος. Η Επίτροπος όταν αναφέρθηκε στην περιφερειοποίηση και την ε, σχέση της, ε, τη σημασία που της δίνεται στην πράσινη βίβλο ήξερε ήδη πώς πρέπει να γίνει βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας επομένως γνώριζε τι θα ισχύει. Οι νομικοί λοιπόν εκτός από το να εντοπίσουν ποιες είναι οι δυσκολίες και οι δυνατότητες ε, να γίνει, να υλοποιηθεί κάτι θα πρέπει να προσπαθήσουν να εξεύρουν και τις κατάλληλες λύσεις ώστε να ανοιχτούν οι κατάλληλες οδοί προς την ε, ε, υλοποίηση της περιφερειοποίησης. Μιλήσατε για δυσκολίες, ε, για πράγματα τα οποία είναι αδύνατα, αλλά δεν παρουσιάστηκαν κάποια μοντέλα περιφερειοποίηση. Η Επίτροπος όμως αναφέρεται σε αυτή την πραγματικότητα συνεχώς και αυτό είναι θετικό στοιχείο. Κατόπιν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει και τα Περιφερειακά Συμβούλια Αλληλείας, όπως ε, ακούσαμε και σήμερα. Τα συμβούλια αυτά θα πρέπει να συμμετέχουν όλο ένα και περισσότερο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να τυχάνουν χάνουν ευρύτερη εκπροσώπηση και φυσικά θα πρέπει να του δίνει τη δυνατότητα να ασκούν πλήρω τα καθήκοντά του. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι η διάκριση μεταξύ ερασιτεχνικής ε, και βιοτεχνικής αλληλείας και του υπόλοιπου στόλου. Σαφώς υπάρχουν διαφορετικές πτυχές. Ε, καταρχάς, ουσιαστική διάκριση μεταξύ βιομηχανικού στόλου και ε, πιο μικρού στόλου και φυσικά τι διαστάσεις υπάρχουν με βάση αυτούς τους δύο στόλους και φυσικά ανάλογη πολιτική. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στον ε, νέο ορισμό αυτών των στόλων, μίλησε για τη διάσταση των σκαφών, για τον αριθμό των μελών του πληρώματος και για, ε, για την ισχύ του κινητήρα. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ε, ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού αλληλευτικού στόλου. Υπάρχουν και άλλα μοντέλα. Το τεχνολογικό επίπεδο του αλληλευτικού σκάφους, ε, το είδος ε, που αλλιεύεται, διότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε πιο εύκολα και μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της αλιείας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διάθεση μεταρρύθμισης επί του θέματος αυτό, η οποία όμως είναι κατεπίγουσα για μας. Τρίτο σημείο, οι ζώνες προστατευόμενης αλίευσης. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των ε, ηχθειοποθεμάτων, κυρίως σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες και πιο εκτεθειμένες. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει οι παρεκκλήσεις που διατυπώνονται στα πλαίσια της κοινής αλληλευτικής πολιτικής να ερμηνεύονται καταλήλως. Επειδή προσφάτως υπήρχε μία μείωση των αλληλευτικών αποθεμάτων, σε σχέση με τις προηγούμενες περιοχές, οι παρεκκλήσεις αυτές ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν. Θα πρέπει οι περιοχές να θεωρούνται ακόμα προστατευόμενες, ίσως και να ενισχυθούν. Παραδείγματος χάρη στις υπερπεριφερειακές περιοχές. Θέλουμε να έχουμε ισορροπημένη διαχείριση των οικοσυστημάτων, ιδίως των πιο ευάλωτων οικοσυστημάτων. Και φυσικά Υπάρχει και το θέμα της οικονομικής υποστήριξης των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν περιοχές αλληλείας οι οποίες ε, θα είναι ε, ενδεδειγμένες για, την, ε, για της μικρής κλίμακας αλληλεία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στόχος που θα διασφαλίσει στην ευρωπαϊκή αλληλεία μία αλληλεία η οποία θα μπορέσει να επιτρέψει στους ανθρώπους αυτούς να ζουν και να βγάζουν τα προστοζή τους από την αλληλεία. Και αυτό μας το επιβεβαίωσε και η Επίτροπος στην ακρόασή της ήδη. Θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε κατάλληλο αποθεματικό ενέργειας για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια, αφού ακούσαμε και την Επίτροπο και την Εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να δώσω το λόγο για τέσσερα λεπτά. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι στο Κοινοβούλιο είμαστε πολύ αυστηροί με το χρόνο σε όλους όσου έχουν ζητήσει το λόγο από τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Θα ξεκινήσω με αλφαβητική σειρά, επομένω. θα ξεκινήσω με την Κύπρο και θα δώσω το λόγο στον κύριο Χατζη Νικόλα, ο οποίος θα μιλήσει εξ ονόματος του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Ελπίζω να μην ε, σκότωσα το όνομά σας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονό ότι παρά τη φιλόδοξη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική το 2002, η έκταση και η ταχύτητα εξέλιξη τη κρίση στον τομέα τη αλληλεία είναι όντω ανησυχητική. Η υπερεκμετάλλευση πολλών αλληλευτικών αποθεμάτων συνεχίζεται. Ο αλληλευτικό στόλο εξακολουθεί να είναι υπερδιογκωμένο. Τα συνδυασμένα αποτελέσματα του πλεονάζοντο αλληλευτικού δυναμικού και των μειωμένων επιπέδων πολλών αποθεμάτων ηχθείων οδηγούν σε μείωση της οικονομικής απόδοσης του τομέα της αλληλείας και σε υποβάθμιση της αποδοτικότητας πολλών αλληλευτικών στόλων. Η κοινή αλληλευτική πολιτική βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Απαιτείται να διαμορφωθεί ένα φιλόδοξο σε περιεχόμενο ισχυρό πλαίσιο για μια ριζοσπαστική εκβάθμιση μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Μια αναθεώρηση που θα επιφέρει μια αλληλεία σύγχρονη, ανταγωνιστική ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσει των καιρών, του περιβάλλοντος και της ποιότητας. Στην αναθεώρηση της κοινής αγροτικής κοινής πολιτικής έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις ελλείψεις του παρελθόντος προκειμένου να αντιστρέψουμε την αρνητική σημερινή κατάσταση που σχετίζεται με το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής αλληλείας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούνται συντονισμένες και ολοκληρωμένες δράσεις και εφαρμογή κοινών κανόνων. Εκτιμώ ότι το πνεύμα συνεργασία που πρέπει να μα διακατέχει για τη συλλογική αντιμετώπιση τη σημερινή κατάσταση υπάρχει. Αυτό εξάλλου κατέδειξε και η πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε με την πράσινη βίβλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω το γεγονό ότι ο ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου τη συνθήκη τη Λισαβόνα αποτελεί κρίσιμη εξέλιξη για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Ο αλληλευτικό τομέα, ένα τομέα που ο πολίτη ζητά αύξηση τη δημοκρατικότητα στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, θα υπόκειται στο εξή τη διαδικασία τη συναπόφαση ω η συνήθι νομοθετική διαδικασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρόλο που ω Κύπρο έχουμε απόψει για όλα τα ζητήματα που αποτελούν του στόχου τη νέα μεταρρύθμιση τη κοινή ελευτική πολιτική, θα σταθώ μόνο σε δύο βασικά ζητήματα που έχουν μεγάλη σημασία για τον κυπριακό αλευτικό τομέα, λαμβάνοντα υπόψη τα ιδιαίτερα εθνικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά του νησιού μα. Σε ό,τι αφορά την παράκτη αλληλεία μικρή κλίμακα, υποστηρίζουμε ένα διαφοροποιημένο καθεστώ διαχείριση που να λαμβάνει υπόψη τι ιδιαιτερότητε των παράκτηων στόλων μικρή κλίμακα και των άκρο απομακρυμένων περιοχών. Παρόλο που η αλληλεία είναι ένα μικρό τομέα τη οικονομία τη Κύπρου, εν τούτη ω κλάδο πρωτογενού παραγωγή, είναι για μα ιδιαίτερα σημαντικό να στηριχθεί και να εξασφαλιστεί το μέλλον του. Ταυτόχρονα τασσόμαστε υπέρ της αύξηση των ποσοστών δημόσιας, κρατικής και κοινωτικής χρηματοδότηση, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική βιωσιμότητα των μικρών στόρων και να διασφαλιστεί η δυναμική της τοπικής οικονομίας και των παράκτιων περιοχών. Σε ό,τι αφορά την υδατοκαλλιέργεια, στηρίζουμε τη θέση ότι η αηφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα στη νέα κοινή αλληλευτική πολιτική. Παράλληλα, θεωρούμε απαραίτητη την απλοποίηση των διαδικασιών για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και την αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργεια. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία των κοινοβουλευτικών συναντήσεων που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεικνύουν αφενό τη θέληση για σύμπραξη και κοινή αντιμετώπιση τη σημερινή πραγματικότητα στον ελευτικό τομέα και αφετέρου την επιθυμία τη Ένωση στα εθνικά κοινοβούλια να έχουν ενεργό ανάμειξη σε ό,τι διαλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το θέμα η ανάδειξη των εθνικών κοινοβουλίων στο κοινοτικό και ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να συνεχιστεί καθώ τα εθνικά κοινοβούλια και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αποτελούν από κοινού τα σημεία σύνδεση των πολιτών με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σα. Να δώσω στη συνέχεια το λόγο στον εκπρόσωπο του Βελγίου από τον Πλάσ Parliament, τον κύριο Κόμπρετ. και να πω ότι ξεκινάει τώρα ε, η διαδικασία να, για να σημειώσετε το όνομά σας στο δεύτερο γύρο. Θα σας διανεμηθούν τα έντυπα τα οποία είναι για το δεύτερο γύρο τώρα. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Dank u wel mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνάντηση αυτή, διότι η πολυπλοκότητα της μεταρρύθμισης της ΚΑΟΠ είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Η αναδιοργάνωση του στόλου δεν είναι το μόνο πρόβλημα, το είπε και η Επίτροπος, πόσα προβλήματα υπάρχουν δηλαδή και η διατήρηση της βιοτεχνικής αλληλείας όσο και η βιωσιμότητα αυτής. Όλα αυτά τα λέει η πράσινη βίβλος βέβαια για, τις τα διαρθρωτικά προγράμματα και τις δημόσιες επενδύσεις ή χρηματοδοτήσεις τους και αφορούν και τη βιώσιμη αλία και την έρευνα αλλά και τον κοινωνικό τομέα, την κοινωνική πτυχή. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να ληφθούν όλα αυτά μαζί υπόψη. Είπατε για τους μικρούς στολίσκους και την βιώσιμη απασχόλησή τους ότι ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα ώστε η μικρή ερασιτεχνική, βιοτεχνική αυτή αλία να διατηρηθεί εμείς ως εκπρόσωποι του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου θα θέλαμε να πούμε ότι η αλληλεία και η εργασία στους λιμένες είναι κύρια δραστηριότητα για πολλές παράκτιες περιοχές της Ένωσης και θα πρέπει να μπορέσει να επιβιώσει και μετά την μεταρρύθμιση που είναι απαραίτητη. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Δανέζικου Φόλκετινγκ, τον κύριο Ντακέλεγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Δανέζικης Βουλής του Φόλκετινγκ σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση της συνάντησης αυτής. Λέγομαι Τελεκιούρτ και εκπροσωπώ τους συντηρητικούς είναι πολύ ευχάριστη για μένα η σημερινή μας συνάντηση γιατί θέλω να εκφράσω τις ανησυχίες μας ως προς την δυνατότητα διατήρησης μιας βιώσιμης αλληλείας. Από το 2009 είχαμε συζητήσει στα πλαίσια της Πρασίνης Βίβλου το θέμα αυτό και φαίνεται ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που μπορούν να λυθούν μόνο αν υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερομένων. Ένα από τα προβλήματα αυτά είναι η υπερβολική αλληλεία, η υπεραλίευση, που αν δεν γίνει κάτι για να αντιμετωπιστεί θα καταλήξει στην εξάντληση όλων των αποθεμάτων και αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις. Το, η μελλοντική κάλπ λοιπόν πρέπει να έχει ως γενικότερο στόχο να εγγυηθεί την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ηλεκτρικής δραστηριότητας καθώς και να τη συνδέσει με διάφορους άλλους τομείς. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να καταλήξουμε στον περιορισμό της υπεραλίευσης και στην απλοποίηση των ελέγχων έτσι ώστε να ωφεληθούν και οι χρήστες και το κοινό. Ο κύριος Μοχλός που προτείνεται είναι μία σειρά κινήτρων ώστε να μειωθούν και οι απορρίψεις και να μην χρειάζονται πια οι ποσοστώσεις. Η ελευθερία επιλογής για την αλληλεία των διαφόρων ειδών θα μπορούσε να καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα εφόσον δίνει στους αλληλείς την ευθύνη να κάνουν την επιλογή. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί αν ο υπάρχον κανονισμός συμπληρωθεί ή αντικατασταθεί ώστε να υπολογίζει ο κάθε αλλιεύς με βάση τα στοιχεία που θα έχουν δοθεί στο παρελθόν τι ευθύνη έχει για την αλλιεύσή του. Έτσι νομίζουμε ότι θα διορθωθούν τα πράγματα και θα υπάρχει μία, για να το πω έτσι, ελεύθερη ποσόστοση. Αυτό θα αποτελούσε με τη σειρά του κίνητρο για να επιλέξουν οι αλληλείς τις καταλληλότερες εγκαταστάσεις και μηχανήματα που να χρησιμοποιήσουν. Ως φυσική επίπτωση της επιλογής του αλλιέως να καταλήξει στο οικονομικά πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Έτσι όμως θα σημαίνει ότι αλλάζει και το σύστημα ελέγχων Πρέπει να υπάρχει επαρκής καταγραφή των αλλιευμάτων ώστε και με τη βοήθεια των δαρυφόρων να είμαστε βέβαιοι για τα στοιχεία που θα διαθέτουμε. Οι κανονισμοί για τα αλλιεύματα πρέπει να συμπληρωθούν από το υπάρχον σύστημα ποσοστώσεων ώστε να μην υπάρχει πια το σύστημα των ποσοστώσεων και κιλοβάτα, αλλά μόνο ποσοστώσεων και αλληλευμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο εκπρόσωπος της Εσθονίας, ο κύριος Μάρκος Σόσαρ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς οι σοσιαλδημοκράτες του, της Εστονικής Βουλής διαβάσαμε σχετικά με την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερος σημαντική. Αλλά επιπρόσθετα προς τις, ε, επιπλέον προς τις άλλες διαστάσεις, άλλες πτυχές, η Αλία παρουσιάζει και μια πολιτιστική διάσταση. Γιατί πολλές, ε, πολλά έθνη που ζουν στη Βαλτική θάλασσα θεωρούν ότι η Αλία είναι αναπόσπαστο, κομμάτι της ε, παράδοσής τους. Ο Γουστάβος ο Τρίτος, ένας Σουηδός βασιλέας, εάν δεν πλανώμε, είπε κάποτε ότι η πίκοή του θεωρούσαν, ε, έτρωγαν τα μικρά ψάρια μαζί με τα κόκαλα γιατί θεωρούσαν ότι είναι πολύ καλά για την υγεία. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σημαντική η κοινή ελευτική πολιτική, αλλά θέλουμε να τονίσουμε κάποιες πτυχές όσον αφορά τη μεταρρύθμισή της μέσω της πράσινης βίβλου. Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό να υποστηρίξουμε τα ITR, R, συγγνώμη, Άρα, Θα πρέπει να υποστηρίξουμε μέσω αυτών την παράκτια αλία γιατί, γιατί η εμπορική αλία πολύ συχνά συγκεντρώνεται στα χέρια ορισμένων μόνο επιχειρήσεων και υπάρχει αυτή η υπερσυγκέντρωση. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διασυνδέσεις μεταξύ των ε, παραγωγών, των αλλιών και των καταναλωτών. Τα μικρά ψάρια είναι ιδιαίτερως φθηνά όταν ε, εκφορτώνονται στην Εσθονία. Αλλά στα καταστήματα είναι ιδιαίτερως ακριβά για τους και αυτό δεν είναι δίκαιο για τους καταναλωτές. Επίσης έχουμε την άποψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει μια συνεργασία με τους ε, αλείς και να συμπεριληφθούν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γιατί οι αλείς θα πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι λαμβάνονται και ήδη υπόψη τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στους επιστημονικούς ε, κύκλους. Και ε, υπάρχουν και πολλές γυναίκες που δουλεύουν σε αυτό το κλάδο στην Εστονία και θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουν στη συζήτηση εν σχέση με την βιώσιμη αλία. Έχουμε, ε, ή μάλλον θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι η αλία είναι μία, ένας από τους τελευταίους παραδοσιακούς τρόπους επιβίωσης για τους ανθρώπους το ψάρι είναι πολύ σημαντική πηγή τροφής. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε, να συγκεντρωθούμε και στις, ε, λεγόμενες, στη λεγόμενη δατοκαλλιέργεια. Γιατί να μην ε, υποστηρίξουμε περισσότερο παραδοσιακούς τρόπους ε, παράκτη αλίας. η πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης εξαρτάται από την αλία μας. Όλες οι παραδόσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαφέρουν μεταξύ τους. Έχω σκεφτεί πάρα πολύ πάνω, πάνω σε αυτό το θέμα. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε τη γλώσσα των ψαριών, ίσως ε, θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε και την ανάγκη να διαφυλάξουμε την βιολογική ποικιλομορφία. Ευχαριστώ. Ε, Στη συνέχεια έχει το λόγο εκ μέρους της ε, Φιλανδίας ο κύριος ε, Μάτις Νίλον για τέσσερα λεπτά. Κυρία Επίτροπε, Αξιότιμοι συνάδελφοι, από την φιλανδική πλευρά είμαστε ιδιαίτερως ευγνώμονες που προσκληθήκαμε σήμερα εδώ σε αυτή την κοινή συνάντηση όπου μπορούμε να συζητήσουμε πολλά σημαντικά θέματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που στην ε, πράσινη βίβλο αναφέρονται τα θέματα της ελίας. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τα, αποθέματα, για τα ληφτικά αποθέματα, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, ε, στις διάφορες ε, περιοχές. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Για μας, το 93% των των από τις ρέγγες αλλιεύονται πριν ε, καν έχουν τη δυνατότητα να αναπαραχθούν. Ε, στην ε, Πράσινη Βίβλο αναφέρονται οι μείζονες γραμμές ελευτικής πολιτικής, αλλά πριν οριστούν θα έπρεπε να συζητηθούν τα θέματα αυτά στο επίπεδο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα για τη Φιλανδία, η παράκτια αλία. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το ζήτημα της ε, αποδοτικότητας και της κερδοφορίας. Ε, πρέπει να ε, υπάρξουν ειδικά αλληλευτικά εργαλεία και για να υπάρξει αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ελής μικρής κλίμακος να έχουν επιδοτήσεις γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει μια βιώσιμη διαχείριση των αλληλευτικών αποθεμάτων εκ μέρους των αλλιέων ε, μικρής ε, κλίμακας. Επίσης το ζήτημα του παροπλισμού των αλληλευτικών σκαφών και εδώ χρειάζεται ε, να γίνει μια προσπάθεια. Χρειαζόμαστε νέα αλληλευτικά σκάφη που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε χωρίς... Ε, να αυξήσουμε το αληφτικό δυναμικό. Και ένα τελευταίο σημείο, οι κανόνες που αφορούν τις επιτρεπόμενες απορρίψεις. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να γίνονται απορρίψεις και ιδιαίτερα στη Βαλτική αυτό είναι πολύ ζημιογόνο ε, και οδηγεί σε μια υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους της ε, Γαλλίας. Καταρχήν, ο εκπρόσωπος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ο κύριος Ντανιέλ Φασκέλ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εμείς ε, είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ μεγάλος βουλευτής, ε, μέλος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και οι συνάδελφοι στη συνέχεια θα παρέμβουν και θα συμπληρώσουν τα όσα θα πω εγώ. Ορισμένα σημαντικά σημεία. Πρώτον, η αναγκαία ενίσχυση της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, ανάγκης ε, να ενημερώνουμε του αλλοί σε σχέση με την ε, μείωση των αποθεμάτων. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν χάσματα μεταξύ των δύο των αλλιέων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν υπάρχει ακριβώς μια διάδοση αυτών των επιστημονικών πληροφοριών. Δεύτερον, εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα των αποθεμάτων με γενικό τρόπο, είναι αναγκαίο να πούμε ναι μεν στην ε, περιφερειοποίηση αλλά ε, γιατί τα θέματα αλίες διαφέρουν από ζώνη σε ζώνη. Εγώ είμαι βουλευτή σε μια περιοχή όπου ε, γίνεται αλία πολλών νυχθείων ταυτόχρονα και, αυτό, και εδώ υπάρχουν πολλές δυσκολίες που θα πρέπει να θέσουμε. Αλλά υπάρχουν άλλοι βουλευτές που μπορούν να αναπτύξουν άλλα θέματα. Άλλο σημαντικό θέμα είναι να συμμετάσχουν οι ίδιοι οι αλλοί στη χάραξη αλληλευτικής πολιτικής. Η περιφερειοποίηση εδώ μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Επίσης η ανάγκη να υπάρχει μια κοινή αλληλευτική πολιτική που να είναι πολυετής γιατί είναι αναγκαίο να υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα. Το να πρέπει να περιμένει κανείς κάθε φορά το τέλο του χρόνου για να ξέρουν οι ΑΕΛΗ πώ μπορούν να λειτουργήσουν και να ζήσουν τον επόμενο έτος είναι αφόρητο για τους ίδιους τους αλληλείς αλλά και για τους επιχειρηματίες και τους μισθωτούς. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη διάσταση. Τώρα όσον αφορά τα ατομικά ε, δικαιώματα νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί εάν κάθε αλληλείας έχει ένα ατομικό δικαίωμα το οποίο μπορεί να μεταφερθεί όπως το επιθυμεί, μπορεί να υπάρξει μια υπερσυγκέντρωση και αποσταθεροποίηση της αλίας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα όσον αφορά την αλία μικρής κλίμακας. Εγώ είμαι υπέρ της άμυνας της αλίας μικρής κλίμακας, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πριν πρόκειται εδώ, γιατί εδώ γίνεται μια συζήτηση αλλά ως το, προς κατόφλι μετά από το οποίο ορίζεται η αλία μικρής κλίμακας ε, μπορεί κανείς ας πούμε να αλλιεύσει την ίδια ποσότητα αλλιευμάτων με λιγότερους ε, αλείς θα πρέπει να προστατεύσουμε την απασχόληση. Ναι, να πούμε ναι στην αλία μικρής κλίμακας που προστατεύει επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επίσης, ε, Επίσης το θέμα των απορρίψεων το οποίο αναφέρθηκε πριν από μένα. Επίσης το ζήτημα των τεχνικών της το οποίο δεν το θέσατε εδώ. Αλλά υπάρχουν τεχνικές αλίες που είναι λιγότερο επιθετικές για το περιβάλλον. Αυτό θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Και επίσης το θέμα των νέων κινητήρων, των υβριδικών ε, κινητήρων νομίζω ότι εδώ θα, εκτιμήσουν οι αλλοί σε αυτού του νέου κινητήρε, αλλά πρέπει να έχουμε την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, πρέπει να ξέρουμε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι διαπραγματεύσει με τι χώρε που δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, το θέμα του Βακαλάου σε σχέση με, τον, με την Ορβηγία μου φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερο ε, σημαντικό και τέλο, θα ήθελα μια κοινή αλληλευτική πολιτική που να, γίνεται πιο, ε, που να είναι πιο εύλογη, να γίνεται πιο εύκολα κατανοητή και να είναι πιο ανθρώπινη. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Γαλλική Γερουσίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στη Γερουσία είναι γνωστό ότι δεν έχουμε στείλει απάντηση στην πράσινη βίβλο της Κομισιόν. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει, αντίθετα μάλιστα γιατί περιμένουμε ακόμη να κάνουμε την πλήρη αξιολόγηση μέχρι να ακούσουμε όλες τις προτάσεις. Θα ήθελα όμως να σας πω ήδη τι συζητιέται στη Γερουσία για τη διαχείριση των πόρων. Υπάρχει το θέμα των μεταβιβάσιμων ατομικών ποσοστώσεων και το είπε και ο συνάδελφος από τη Γαλλική Βουλή. Όλοι μπορεί να συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αναθεώρηση, αλλά καλύτερο θα ήταν πρώτα να γνωρίζουμε ποιοι έχουν δικαίωμα αγοράς ποσοστώσεων, γιατί υπάρχει τεράστιος κίνδυνος συγκέντρωσης κερδοσκόπων. Άλλο θέμα η διαχείριση των απορρίψεων. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να καταστεί εκρηκτικό στο μέλλον. Η λύση όμως δεν θα είναι απλή. Είναι θα ήταν εύκολο να λυθεί αν ήταν σίγουρες οι τοποθεσίες των αποθεμάτων, αλλά όταν πρόκειται για ψάρια του βυθού τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Οι έλεγχοι είναι πολύ δύσκολο να επιβληθούν το ξέρουμε αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε κάποια συνέπειά τους. Τέτοια συνέπεια των ελέγχων υπάρχει, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε εκτός των συνόρων μας. Ερωτώ, μήπως θα μπορούσε να υπάρξει κάποια ετικετοποίηση, για να το πω έτσι, της αλληλίας, ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι η αλληλεία ευρωπαϊκής προέλευσης. Τώρα για το μέλλον της ΚΑΛΠ ποια είναι τα κύρια μαθήματα που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Τρία. Πρώτον, να προσέξουμε μήπως υπάρχει υπερβολική διαχείριση και γραφειοκρατία όπως σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Διότι μια πολιτική που επιβάλλεται εκ των άνω δεν θα γίνει δεκτή. Νομίζω ότι αυτό το μάθημα το δέχονται όλοι. Δεύτερον, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανένα πρόγραμμα αν δεν υπάρχει ανάλογη πολιτική θέληση. Και γι' αυτό θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την κοινωνική πτυχή του προβλήματος. την πτυχή αυτή την έχει κάπως αγνοήσει η Κομισιόν και θα θέλαμε να την προσέξει. Από δύο απόψεις. Μία την επαγγελματική εκπαίδευση του προσωπικού και δύο την ασφάλεια. Γνωρίζετε όλοι και όλες ότι πρόκειται για πολύ επικίνδυνο επάγγελμα. Τρίτο, η σύνδεση που θεωρούμε ότι υπάρχει, η σχέση μεταξύ της ΚΑΛΠ αυτής και της ΚΑΠ διότι η αλία μάλλον θα μεταρρυθμιστεί πριν από την ΚΑΠ και θα θέλαμε όλος ιδιαιτέρως το είπε και κάποιος συνάδελφος από κάποια άλλη χώρα να γνωρίζουμε ποια περιθώρια υπάρχουν στην πράσινη βίβλο λέει ένα κομμάτι κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την οργάνωση των παραγωγών για την αλληλεία προς πώληση. Πρόκειται για εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων και αυτό μας ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερως. Σας κατευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Γερμανίας από τον Bundesrat. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Χαίρομαι πολύ σήμερα που ως εκπρόσωπος του της Γερμανικής Βουλής να σας παρουσιάσω τις απόψεις για την κοινή αλληλευτική πολιτική από την πλευρά όλων των βόρειων ε, ομόσπονδων παράκτιων κρατηδίων. Στην Βόρεια Ριτανία Βεσφαλία έχουμε μια εκτεταμένη συζήτηση ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και έκανα μια τέτοια συζήτηση πριν από μερικού μήνε. Η διάφραση του στόλου μα στα βόρεια ομόσπονδα κρατήδια βασίζεται σε οικογενειακέ επιχειρησιακέ μονάδε. Πρόκειται για αλία μικρή κλίμακα και υπάρχουν, για παράδειγμα, υπάρχει ένα στόλο 77 ληφτικών ε, σκαφών που είναι περίπου 27 μέτρα μήκος. Οι οικογενειακές αυτές επιχειρήσει επιχειρήσεις δημιουργούν πολλές ανησυχίες γιατί η οικογενειακή τους κατάσταση είναι αρκετά δεινή και αυτό σχετίζεται με το υψηλό κόστος που προέρχεται από το υπερβολικό γραφειοκρατικό άχθος. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την αλία και αυτές οι πολυάριθμες νομοθετικές διατάξεις δεν, ε, είναι, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Συνεπώ λοιπόν στη μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να υπάρξουν απτές βελτιώσει στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Θα πρέπει, γιατί ε, μόνο νέε διατάξει από μόνε του δεν αρκούν. Η ΚΑΛΤ θα πρέπει να είναι απλούστερη, διαφανέστερη και συνεπώ πιο εφαρμόσιμη. Οι υφιστάμενε διατάξει θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο βασικός λόγος της αποτυχίας μέχρι τώρα της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Σε όλες τις χώρες μέλη θα πρέπει να υπάρξουν ίδιες προϋποθέσεις ε, πλαίσιο για, τις, ε, για την περίπτωση παραβιάσεων. Τώρα, όσον αφορά την πλεονάζουσα αλία, μέχρι στιγμής ε, δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη το θέμα αυτό στη Γερμανία κατανομή των αλλιευμάτων βάσει τη αρχής τη σχετική σταθερότητα και το σύστημα των εθνικών ποσοστώσεων θα πρέπει να παραμείνουν πυλώνε της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Το ισχύον σύστημα ποσοστώσεων ε, εξασφαλίζει στους ελέγχους ότι οι χώρες παραμένουν συνυπεύθυνες για μια βιώσιμη πολιτική και η Ευρωπαϊκή αλία σε όλες τις παράκτιες χώρες έχει ένα αξιόπιστο μέλλον. Όσον αφορά την ε, τήρηση των κανόνων, είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκές ε, χώρες να είναι συνυπεύθυνες και για τη διαχείριση της πολιτικής αλίας. Γιατί αν πάψει να ισχύει αυτό το σύστημα, η παραδοσιακή παράκτη αλία δεν πρόκειται να επιβιώσει. Όσον αφορά τώρα τη βιωσιμότητα της αλίας μικρής κλίμακας θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου η δυνατότητα επιδοτήσεων βεβαίως ε, κάτω από την άποψη της εξασφάλισης των θέσεων εργασίας. Βεβαίως η βιώσιμη διαχείριση των πόρων θα πρέπει να παραμείνει πρώτη στο στόχο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και εδώ εντάσσεται ε, ε, το θέμα των απορρίψεων ε, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί μια τελική ε, λύση. Και ένα άλλο ρέθισμα. Ε, στην Βαλτική έχουμε, το ειδικό, έχουμε πολύ ειδικά προβλήματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ορθό να δούμε πώς μπορεί κανείς με την ενίσχυση των περιφερειακών γνωμοδοτικών οργάνων να ενισχυθούν οι περιφέρειες. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της γραφειοκρατίας και σε ε, επιβάρυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ναι, ευχαριστώ πολύ την κυρία Γρούμφ. Από Γερμανία και πάλι, αλλά από τον Bundestag. Ε, κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι ε, συνάδελφοι, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή πρόσκληση. Ε, εγώ είμαι πολιτικός εδώ και 15 ε, χρόνια, γι' αυτό δεν θέλω να λειτουργήσω μόνο διακοσμητικά. Ε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Τα περιφερειακά, όσον αφορά τα περιφερειακά όργανα, εμείς έχουμε κάτι ανάλογο στην Βόρεια Θάλασσα. Ένα τρίτο των μελών που βρίσκονται εκεί, που συμμετέχουν εκεί, συγγνώμη, είναι μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και αυτό λειτουργεί εξαιρετικά. Μόνο που έχω την αίσθηση και πολύ συχνά έχω και τις αποδείξεις ότι αυτό που ε, γίνεται εκεί αντικείμενο επεξεργασίας δεν λαμβάνεται υπόψη στις Βρυξέλλες ποιος ε, λέτε ότι, λέτε ότι είστε υπέρ των περιφερειακών ε, συμβουλίων, αλλά τελικά η δουλειά τους παραμένει στα συρτάρια. Τώρα, όσον αφορά την ε, παράνομη αλία, ε, είπε κάποια πράγματα κυρία Ρούμφ. Λέτε κυρία Επίτροπε ότι θέλετε να ενισχύσετε την αλία μικρής ε, κλίμακας. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό δείγμα. Χρειαζόμαστε υποστήριξη, ωστόσο, για την, τον εξυγχρονισμό του στόλου. Ο γερμανικός στόλος είναι πάνω από 30 ετών, τα σκάφη είναι πεπαλαιωμένα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, την ασφάλειά τους. Δεν είναι δυνατόν όταν η αλλιέας θέλει να βάλει ένα νέο κινητήρα, αναφέρθηκε από το παράδειγμα του υβριδικού μοντέλου, ε, ε, και στη συνέχεια έχει 25% επιδότηση αλλά αυτός πρέπει να δώσει 50% ε, του κέρδους για τον κινητήρα. Μιλήσατε επίσης για την ε, κατασπατάληση του αποθέματος για την εξάρτηση του αποθέματος. Αλλά δείτε τι, τι έκαναν οι προκάτοχοί σας. Είχαμε στις ε, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα την εντολή των απορρίψεων και με τα, μικρότερα διάκαινα ήταν ε, περισσότερες οι απορρίψεις από ό,τι με τα μεγαλύτερα διάκαινα των ε, δικτυών. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να επίσης να δώσουμε περισσότερα κονδύλια για την έρευνα. Θεωρώ κυρία Επίτροπε ότι ξέρετε και αυτό δεν μπορεί να ότι στη Γερμανία δεν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός αλληλευτικός στόλος. Υπάρχουν μόνο εθνικοί στόλοι. Εάν ε, προσθέσουμε το δυναμικό των ευρωπαϊκών χωρών, θα διαπιστώσουμε ότι στη Γερμανία ε, είναι ε, μόνο το 3% του συνολικού αλληλευτικού, της συνολικής αλληλευτικής ικανότητας. Τώρα, όπως για τα παρεπέμπτοντα αλληλεύματα, θα πρέπει να φροντίσετε αυτό. Θεωρώ ότι είναι καλό όταν διατηρήσουμε μια σχετική σταθερότητα και θα ήθελα να σας υποστηρίξω εάν πράγματι είναι αυτή η άποψή σας και οι εθνικές ποσοστώσεις θα πρέπει να μπορούν να αλλάξουν, αλλά όχι να γίνονται αντικείμενο εμπορίας. Γιατί ε, δεν είναι δυνατόν να υποφελούνται μόνο όσοι έχουν τα χρήματα. Έτσι ζημιώνονται οι διαλύσεις. Τώρα, όσον αφορά την αλλία μικρής κλίμακας. Ε, πώς τη μετράμε βάσει του μήκους των αλληλευτικών σκαφών. Τώρα, όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες, εκτός της Ευρώπης, στις υδατοκαλλιέργειες υπάρχουν ε, διψήφια, διψήφια αριθμοί ανάπτυξης. Όχι όμως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα ήθελα, κυρία Επίτροπη, να συζητήσετε με τους συναντάλφους σας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Τονίστηκε η σημασία της παράκτης αλίας. Στη Γερμανία ε, ψαρεύονται ένα έβδομο των ε, ψαριών που χρειάζονται. Τα υπόλοιπα ψάρια εισάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες. Στη Γερμανία έχουμε περίπου 30-35 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ε, στην Αλία έχουμε 43.000 μόνο. Η θέση απασχόληση δεν είναι το ισχυρότερο επιχείρημα. Το ισχυρότερο επιχείρημα ε, προήλθε από, το, από την ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης όπου ελέγχθη ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας η Αλία. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω, πρώτο δεκίβημα είναι η ταυτότητα των ακτών μας, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Δανία, είτε στη Λιθουανία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Από πλευράς Ελλάδος τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μιχαήλ Τσελέπης για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ελλάδα συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη μεταρρύθμιση της κοινή αγρο... αλληλευτικής πολιτικής και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία για να επιτύχει τους στόχους της τόσο σε επίπεδο της κατάστασης των απεθυμάτων όσο και στη βιωσιμότητα της αλληλείας και της οικονομικής κατάστασης του τομέα. Η βασική άξονε στου οποίου η μελλοντική κοινή αλλιευτική πολιτική πρέπει να στηριχθεί σύμφωνα με τη χώρα μα είναι η διασφάλιση τη προοπτική του ευρωπαϊκού αλλιευτικού τομέα και τη ικανότητα προσαρμογή του στι νέε ανάγκε που δημιουργούνται αφενό από την ανεπάρκεια των πόρων και αφετέρου από τη ζήτηση τη αγορά σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίηση τη και αύξηση του ανταγωνισμού. Η διασφάλιση τη αηφορία των αλλιευτικών πηγών υιοθέτηση απλών δίκαιων και εφαρμόσιμων αρχών ώστε η μελλοντική κοινή αλλιευτική πολιτική να είναι αποδεκτή από εκείνου του οποίου αφορά. Η έμφαση στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση του τομέα ώστε να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπέ επίπεδο διαβίωση για του αλληλεί. Η έμφαση στην ασφάλεια και στην εργασία. Η οικονομική στήριξη του τομέα για την προσαρμογή του στου στόχου τη μελλοντική κοινή αλληλευτική πολιτική. Όσον αφορά τη Μεσόγειο, η διαχείριση της αλληλευτικής προσπάθειας εν μέσω διαχείρισης των πόρων και της αλληλείας πρέπει να παραμείνει σύμφωνα και με τους προσανατολισμούς της Γενικής Επιτροπής Αλληλείας της Μεσογείου. Στη Μεσόγειο η διαχείριση των πόρων δεν μπορεί να στηριχθεί στο εργαλείο των συνολικά επιτροπόμενων αλλιευμάτων και στον προσδιορισμό της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, καθώς η αλληλεία είναι πολυειδική και, και περισσότερα είδη στοχεύονται από πολλά αλλιευτικά σκάφη βασικό εργαλείο διαχείριση των πόρων στη Μεσόγειο πρέπει να είναι η εφαρμογή τεχνικών μέτρων και η αύξηση τη επιλεκτικότητα των αλλιευτικών εργαλείων προκειμένου να ελαστικοποιηθούν οι απορρίψει. Με αυτόν τον τρόπο υπηρετείται ο στόχο των μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων. Για την παράκτη αλία η διαχείριση αυτής της δραστηριότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την κοινή αλληλευτική πολιτική με ιδιαίτερο τρόπο με βάση τα χαρακτηριστικά του στόλου που την ασκεί των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μεσογείου στην οποία ασκείται όσον αφορά την ελληνική αλληλεία και τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών που εξαρτώνται από αυτήν στα οποία μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ιδέουσα σημασία. Η διαχείριση της παράκτιας αλληλείας είναι ανάγκη να διαφοροποιηθεί από τη διαχείριση της βιομηχανικής αλληλείας. Όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες, η χώρα μας υποστηρίζει ότι ο τομέα των υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της νέας κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας ανεξαρτήτως μεγέθους αλλά με γνώμονα τη συμβολή του στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της στασιμότητας της παραγωγής που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργεί ένα ελληματικό εμπορικό ισοζύγιο λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Για το εμπόριο και αγορές θα ήθελα να προσθέσω ότι στο πλαίσιο της νέας κοινή αλληλευτικής πολιτικής και όσον αφορά τον τομέα της εμπορίας και των αγορών θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι βασικές αρχές που διέπουν τον εφοδιασμό των αγορών με ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και τη συμμετοχή των παραγωγών στην εμπορία της παραγωγής τους και η κοινή αλλιευτική πολιτική κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της αλληλείας την οποία έχει υποτιμήσει σε σχέση με την περιβαλλοντική και οικονομική. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί προκειμένου να προσφέρει ουσιαστική στήριξη ιδίω σε περιοχέ που ο τομέα διαδραματίζει έναν πλέον δυναμικό ρόλο προσφέροντα ουσιαστικά κίνητρα εισαγωγή νέων στο επάγγελμα του αλληλεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά Ιρλανδίας τώρα έχουμε δύο εκπροσώπους των δύο βουλών αντιστέχων. Καταρχά ο κύριο Τόμ Σίχαν, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι η πρόσβαση και για να αντιστρέψω το σχόλιο της Επιτρόπου για τα ITQ νωρίτερα, η Ιρλανδία προτείνει η πρόσβαση στα παράκτια είδητα να εξεταστεί και να επεκταθούν ε, τα χωρικά είδατα στα 20 μίλια με συγκεκριμένες ρυθμίσεις ε, για να βοηθήσουμε τις ε, συγκεκριμένες κοινότητες που εξαρτώνται από την παράκτια ηλία. Η Ιρλανδία φρονεί ότι τα ε, χωρικά ύδατα των κρατών μελών θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο για αλίευση από τους ε, κατοίκους της χώρας και να λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη ιδιαίτερη κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η πρόσφαση στα παράκτια είδετα ε, είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό πρόβλημα για τους αλληλείς και έχουν γίνει πολλές συνεδριάσεις στη χώρα κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Γι' αυτό και η Ιρλανδία θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω παράταση ε, στην ε, επέκταση στα χωρικά ύδατα και να έχουμε 20 μίλια και τα 6 μίλια να επεκταθούν στα 10 μίλια και η περιοχή 6-12 μιλίων να γίνει 10-20 μιλίων. Επιπλέον, τα παράκτια ύδατα είναι φυσική οικοτοπή για γόνους ψαριών και για πολλά είδη οστράκων. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πολλές ανθρώπινες επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η μόλυνση των ακτών και ο τουρισμός που ε, παρεμποδίζουν αυτές τις δραστηριότητες. Γι' αυτό λοιπόν οι πιο ανεπτυγμένε ε, χώρες των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των παράκτιων περιοχών και να έχει μία προσέγγιση που θα σέβεται το οικοσύστημα. Η Ιρλανδία θα ήθελε οι αυτόχθονες νησιωτικές κοινότητες όπως αυτές που έχουμε στις δυτικές ακτές της Ιρλανδίας να υποστηριχθούν για να αναπτυχθούν προγράμματα αλίας από την οποία εξαρτώνται. Το άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να θέξω είναι η υδατοκαλλιέργεια. Η Ιρλανδία θέλει ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής Ιδετοκολοέργειας με έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα καθορίζει μια πορεία αυξανόμενης αρμονίας με κοινοτικούς περιβαλλοντικούς νόμους πιστεύετε ότι η ζήτηση για τα θαλασσινά θα συνεχίσει να αυξάνεται και επομένως δεν θα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές μόνο με την ε, ε ηχθειοκαλλιέργεια ε, η οποία γίνεται σε ε, ελεύθερα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η δατοκαλλιέργεια. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αποφύγουμε τα εισαγόμενα προϊόντα διότι αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των, προϊό... τροφίμων και να προτιμήσουμε τα ενδοκινοτικά προϊόντα. Επομένως θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η υδατοκαλλιέργεια. Η Ιρλανδία παρέχει πολλά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και θεωρείται ότι θα μπορούσε να έχει μια αύξηση κατά 60% μέχρι το 2020. Υπάρχει πίεση για τις αγορές ε, προϊόντων αυτών και υπάρχουν και πολλές ε, ε, Ανησυχίε για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του κλάδου. Και επομένω θα πρέπει να ληφθούν μέτρα περί αυτού. Θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα ε, τα οποία θα βοηθούν την ανάπτυξη της αλληλεία ε, αλληλείας ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος. Η υδατοκαλλιέργεια είναι σημαντική και για την διατροφική ασφάλεια αλλά και για να μπορέσει να καλυφθεί το έλλειμμα πληρωμών που προκύπτει ακριβώς από την υπερβολική εξάρτηση από εισαγόμενα αλλιευτικά προϊόντα. Θεωρούμε ότι η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί και όχημα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ και τώρα από πλευράς ε, Ιρλανδικής Γερουσίας ο κύριος Μάικολ Μακάρθη. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Συνάδελφοι, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ από πλευρά Ιρλανδικού Κοινοβουλίου για να παρουσιάσω τη θέση της Ιρλανδία για τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής ε, πολιτικής. Θα ήθελα να σταθώ στα ITQs, την αρχή της σχετικής σταθερότητας, τις προτιμήσεις και το θέμα των απορρίψεων. Στο Συμβούλιο Αλληλείας οι Υπουργοί καθόρισαν τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα για το 2010 και αυτά βασίζονται στα ιστορικά στοιχεία που έχουμε και το λαμβάνοντας υπόψη και το στοιχείο της σχετικής σταθερότητας. Τα κράτη-μέλη καθορίζουν πώς δίνονται οι ποσοστάσεις μεταξύ αλλιέων. Στην Ιρλανδία αυτή η διαδικασία θεωρείται δημόσιο αγαθό. Mm. Είμαστε ιδεολογικά αντίθετοι λοιπόν στο θέμα της ιδιωτικοποίησης και κάνω έκκληση προς εσάς κυρία Επίτροπε να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα και να διατηρήσετε αυτή την κατάσταση ε, προς όφελος των αγροτικών και παράκτιων ε, οικονομιών ανά τον κόσμο και κυρίως για την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία προσπαθεί να καταπολεμήσει την ύφεση όπως και πάρα πολλές άλλες χώρες και αυτός είναι ένας από τους τομείς που μας έχουν γονατίσει. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να σταματήσουμε, να ανακόψουμε αυτή την τάση, να έχουμε ένα ε, πλαίσιο το οποίο είναι ουδέτερο από πλευρά εισοδήμων και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τι κοινότητε που βασίζονται στι θαλάσσιε δραστηριότητε. Γι' αυτό ακριβώ κάνω έκκληση προ εσά, κύριε Επίτροπε να δείτε τι κοινωνικο οικονομικέ υποπτώσει αυτή τη διαδικασία και να επιτρέψετε να παραμείνει η κατάσταση ω έχει. Για την Ιρλανδία η παράκτη αλληλεία είναι εθνικό αγαθό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει εθνικό αγαθό. Αν επιτραπεί να προχωρήσουν οι θέσεις ε, άλλων κρατών μελών που είναι αντίθετες προς τη δική μας, ε, θα υπάρχει πρόβλημα, δεν θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν οι ποσοστάσεις, θα πρέπει να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο και να κατανέμονται ως εθνικό αγαθό. Θα πρέπει να κατανοήσετε πόσο σημαντικές είναι οι ε, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις για μας, κύριε Επίτροπε. Επίσης, θεωρούμε ότι το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι δίκαιο σύστημα και στα πλαίσια τη κοινή αλληλευτικής πολιτικής ζητούμε να παραμείνει ως έχει είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμά να κατανοήσουμε την άποψη άλλων κρατών μελών για το θέμα της σχετικής σταθερότητα. και θεωρούμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγχουμε τα τάκ αυτό είναι το πιο δίκαιο σύστημα και ε, ορισμένες φορές υπάρχουν κάποια συμπληρωματικά μέτρα μεν, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει η κατάσταση ως έχει, όπως είπα και πριν. Στην ε, Συμφωνία της Χάγης του 1956, αν ανακληθεί, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δοθούν επιπλέον ποσοστάσεις. Η συμφωνία αυτή δημιουργήθηκε ακριβώς για να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η Ιρλανδία είχε υποανεπτυγμένη αλληλευτική δραστηριότητα το 1996 όταν εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προστατεύσουμε τις παράκτιες περιοχές, ε, ο πληθυσμός των οποίων εξαρτάται από την αλληλεία και θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε μια προστατευόμενη περιοχή αλίας. Τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα μας και θεωρούμε ότι το σύστημα αντικατοπτρίζει μια πολύ σημαντική πολιτική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών μας και ζητούμε όχι μόνο να παραμείνει το status quo, παρά Επίσης ζητούμε να παραμείνουν οι προτιμήσεις ε, του συστήματος της Χάγης ε, και στο μελλοντικό σύστημα. Αυτή είναι η θέση μας και ελπίζω να καταλάβετε για ποιον ακριβώς το λόγο ε, την υποστηρίζουμε. Τώρα, για το θέμα των απορρίψεων. Ξέρουμε ότι αυτό το θέμα είναι διαφιλονικούμενο και ε, θέλουμε να υπάρχει απαγόρευση απορρίψεων για αποθέματα τα οποία πραγματικά πλήττονται θα θέλαμε να αλλάξουν πρακτικές για να μειωθούν τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα τα οποία είναι επιθύματα, τα οποία θα πρέπει να γίνονται σε συνδυασμό με τη βιομηχανία, τους επιστήμονες ε, και τους αλληλείς για να μπορέσουμε να βρούμε ποια είναι τα συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθηθούν περισσότερο. Κάνω έκκληση κύριε Επίτροπε να δούμε τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ από την Ιταλική Βουλή ο κύριος Πάουλε Ρούσι Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ γιατί είναι πολύ επίκαιρη αυτή η δυνατότητα που μας δίνεται να συζητήσουμε μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Η κοινή αλληλευτική ε, πολιτική βρίσκεται ενώπιον μιας ε, συγκυριακής κρίτησης και υπάρχουν ε, μη ικανοποιητικά αποτελέσματα στις κοινοτικέ πολιτικές αλληλείας. Δεν λαμβάνει μέρευμα για τα θέματα της εργασίας και της αξίας της βιωσιμότητας και της ισορροπίας του περιβάλλοντος. Η βιολογική κατάσταση των ηχθειοποθεμάτων δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά, κυρίως λόγω της αλλιευτικής ικανότητας του στόλου των κρατών μελών, η οποία είναι ακόμα υπερβολική σε σχέση με τα θαλάσσια αποθέματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης και η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων δεν έχει βελτιωθεί και το θέμα της απασχόλησης είναι σε συνεχή μείωση. Η κρίση του καυσίμου του 2008 ε, δημιούργησε μια πιο διαρθρωτική δυσκολία. Κατά το διάστημα 2004-2008 στην Ιταλία χάθηκαν περίπου 5.500 θέσεις εργασίας. Ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια μεταρρύθμιση, αλλά μια εκβάθρον μεταρρύθμιση που θα αλλάξει ε, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή προσφέρει μεγάλο άχθος, είναι πολύ περίπλοκο και ορισμένες φορές μπορούμε να πούμε ότι είναι και προτιμησιακό. Θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια μορφή επικουρικότητα. Ένα κέντρο το οποίο θα αποφασίζει και θα δίνει τις κατευθύνσεις και μια περιφέρεια που σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα καθορίζει τους κανόνες υλοποίησης και θα τους θεωρεί δικούς τους. Επομένως θα συμμετέχει. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε τους τοπικείς φορείς και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να αναπτυχθεί η πραγματική τους οικονομική αξία. Μόνο αν έχουμε βιώσιμη αλληλεία μακροπρόθεσμα μπορούμε να έχουμε ένα οικονομικό μέλλον ε, εισάξιο του τομέα αλλά φυσικά η οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται αποκλειστικά από τη διατήρηση των αποθεμάτων. Επομένως η Ευρώπη θα πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο για να μπορέσει να καταπολεμήσει ακόμα περισσότερο, με περισσότερο σθένος και περισσότερο θάρρος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την παράνομη, άναθρη και λαθρέα λία. εν τέλει θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, κατά την άποψή μου, τη δυνατότητα να έχουμε στοιχεία περιφερειακής ανάπτυξης για να μην έχουμε πολύ αυστηρή κεντρική ε, διαχείριση ε, και πολύ υπερβολική κεντρική διαχείριση θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση για τη μικρή κλίμακα η οποία μπορεί να διαδερματίσει ουσιαστικό ρόλο για την οικονομική βιωσιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του κάθε χώρου ω αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής και περιβαλλοντικής κατάστασής του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ρούσο. Από την Πολωνία τώρα, από πλευράς Γερουσίας. Ο κύριος Κροτσικόφσκι. Ελπίζω να μην το πρόφερα πολύ άσχημα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Μιλώ εξ ονόματος της Πολωνικής Γερουσίας Και θα ήθελα να σας πω ότι θεωρούμε ότι υπάρχουν ορισμένα σημαντικά προβλήματα που πρέπει να θυγούν εδώ. Είναι σημαντικό, αφού συζητάμε την κάλπα, να αναγνωρίσουμε ότι ακούγονται πολλές και πολλαπλές φωνές και διαφορετικές απόψεις και είναι σημαντικό να τις δούμε όλες. Όλοι μας θέλουμε να υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποια μεταρρύθμιση, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή βιώσιμη ανάπτυξη και να διασφαλιστεί το μέλλον της αλίας. Οι αλληλείς και τα αλλιευτικά πλοιάρια λοιπόν πρέπει να διατηρηθούν, να υπά... συνεχίσει να υπάρχει μια ισορροπία έτσι ώστε το, τα έσοδα των αλλιέων να παραμείνουν σε αποδεκτό επίπεδο. Το κλειδί εδώ είναι ίσως να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής αλληλείας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ακόμη εισάγουμε ψάρια και δεν πρέπει να δούμε την Ένωση σε απομόνωση με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να διασφαλίσουμε βέβαια και την ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια για τα αλλιευτικά προϊόντα ώστε να γνωρίζουμε ανα πάσα στιγμή την προέλευσή τους. Είναι προφανές ότι η αλληλεία δεν είναι η μόνη διάσταση της τοπικής οικονομίας, είναι ένα τμήμα ενός ολόκληρου δικτύου τοπικής οικονομίας αλλά ο τομέας αυτός είναι πάντοτε σημαντικός τοπικά και πρέπει να μπορέσει να διατηρηθεί. Η αποκέντρωση λοιπόν και η περιφερειοποίηση καθώς και η απλοποιημένη διαχείριση θα είναι αποφασιστικά στοιχεία για τη μεταρρύθμιση αυτή και αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος, να υπάρχει καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Αυτά ακούσαμε και σήμερα από την κυρία Επίτροπο οι μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις, μεταφέρσιμες ποσοστώσεις είναι και αυτές ε, τμήμα της λύσης αλλά όπως είπε και κάποιος προηγούμενος ομιλητής υπάρχουν και φόβοι επί όλων αυτών για τις απορρίψεις και την υπεραλίευση νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συνεχιστούν πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι απορρίψει θα ελεγχθούν τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Αλία, ιδιαίτερα δε στη Βαλτική. Γιατί αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης και βιώσιμης διατήρησης μάλιστα των αποθεμάτων μας. Πρέπει να δούμε πώς ήταν η κατάσταση, να κάνουμε μια αναθεώρηση, μια να έχουμε μια εποπτεία της ιστορίας όλων αυτών των πραγμάτων και ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς και η μόνη των εθνικών βουλευτών. Ωραία. Ο κύριος Λάντης Λαβλούκα πάλι από την Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία και κύριοι βουλευτές θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τέσσερα προβλήματα που σχετίζονται με την ΚΑΟ. Γενικά η Πολωνία υποστηρίζει το σκεπτικό που ακούστηκε και σήμερα ότι την αναγκαιότητα δηλαδή για αναθεώρηση της ΚΑΛΠ, για μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ. Συμφωνούμε με την Επιτροπή, με την Κομισιόν ότι πρέπει η κατάσταση της αλίας να βελτιωθεί, της αλιευτικής βιομηχανίας Έχουμε ορισμένα εργαλεία, υπάρχουν τα αλληλευτικά ταμεία και είναι κάτι που δεν, ε, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, δεν είναι αμεληταίο. Πρέπει να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη χρησιμοποίηση των υπάρχοντων χρημάτων για την σωστότερη δυνατή κατανομή τους. Πιστεύω ότι το 1 τρίτο του αλληλευτικού μας στόλου έχει χαθεί, έχει απολεστεί. Ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Το 1 τρίτο του στόλου μας, επαναλαμβάνω, έχει απολεστεί, έχει χαθεί, έχει μειωθεί. Πρέπει απαραίτητος να γίνει μια μεταρρύθμιση αλλά ρεαλιστική και αξιόπιστη Γι' αυτό μιλάμε μάλλον για περιφερειοποίηση και αποκέντρωση. Γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ακριβή επιστημονική πληροφόρηση που να συνοδεύει την περιφερειοποίηση, δηλαδή μια νέα διαδικασία λήψης αποφάσεων και συντονισμού μεταξύ Βρυξελών και περιφέρειας και η ΚΑΛΠ δεν πρόκειται να πετύχει παρά μόνο να υπάρξει αναδιάρθρωση και των χρηματικών της. Πρέπει να, υπάρχει σαφής, να υπάρχουν σαφείς και διαφανείς αρχές για τη διαχείρισή της. Να δούμε και ποιες είναι οι ευχές και οι πόθη των ίδιων των αλλιέων. Το κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια φυσικά το ξέρουν αυτό, το βλέπουν ε, σαφώς, καθαρά. Γιατί είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ζωή των κατοίκων των παρακτήων περιοχών. Και τώρα για να τελειώσω θα ήθελα να δείξω ένα μόνο ακόμη θέμα σχετική σταθερότητα. Εμείς είμαστε υπέρ της διατήρησης της αρχής αυτής της σχετικής σταθερότητας με τη μορφή που έχει σήμερα. Γιατί είναι κάτι βασικό για την κάλπα από την αρχή της. Είναι μια αρχή που έχει αποδείξει την αξία της και κατ' εμάς είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να διατηρηθεί ως ένα από τους πυλώνες της ΚΑΛΠ. Το να αλλάξει η αρχή αυτή νομίζω θα μας ζημιώσει τελικά και θα βλάψει όλο το μέλλον του τομέα. Ο κύριος Οδυσσεύς Περέιρα από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι από τα κοινοβούλια ε, και σας ε, κυρία Νέδες, θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την έκθεσή σας που έτυχε πλατιάς υποστήριξη εδώ στο Κοινοβούλιο. Και το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο ασχολείται εντατικά με αυτή τη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και υπάρχει και μία πλατιά συνένεση σε όλες τις ε, πολιτικές ε, ομάδες. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ε, και υπάρχει μία υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία θα ήθελα να θέσω και τα οποία θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς. Καταρχήν είναι θεμελιώδης σημασία να συνδέσουμε τις τρεις ε, διαστάσεις που καλύπτει η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ε, τα περιβαλλοντικά θέματα, δηλαδή τη διατήρηση των αποθεμάτων και βιωσιμότητα. Ο κοινωνικός ε, πυλώνας για την συνοχή και την αξιοπρέπεια των αλληλευτικών κοινοτήτων. Και επίσης η οικονομική διάσταση, γιατί εάν η αλία δεν είναι κερδοφόρα θα υπάρξουν νέες επενδύσεις. Μία νέα πολιτική λοιπόν θα πρέπει να περιλαμβάνει τις νέες δεσμεύσεις και την αναγκαία υποστήριξη. Δεν θα πρέπει να δώσουμε μία προτεραιότητα στον ένα τομέα και να παραπελήσουμε τους άλλους. Παρά τις ε, προϋποθέσεις που θέτει η νέα συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να κάνουμε κάτι όσον αφορά την ακραία, ε, τον ακραίο συγκεντρωτισμό του ισχύοντος μοντέλου. Θα πρέπει να έχουμε μια κατάλληλη περιφερειακή διαχείριση για να μπορεί να συμμετάσχει και το Κοινοβούλιο στην εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν συνέργεια και ένα κοινό όραμα για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων. Επίσης θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να διορθώνει τις ανισορροπίες στο παρόν σύστημα τόσο όσον αφορά την επιτρεπόμενη αλία στα χωρικά ύδατα των 12 μιλίων καθώς και συζήτηση εν σχέση με τη βιομηχανική αλία. Όσον αφορά τα αλληλευτικά αποθέματα θα πρέπει να έχουμε επαρκείς γνώσεις ως βάση της δημόσιας συζήτησης οι ποσοστώσεις θα πρέπει να εστιάσουν ε, στις ατομικές ε, περιπτώσεις. Ε, όσον αφορά δε ε, τα ατομικά δικαιώματα, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την αλία μικρής κλίμακας. Θα πρέπει κατά άποψή να υπάρχει ένα εκούσιο σύστημα των ITR, ούτως ώστε οι πλειοκτήτες να μπορούν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους εδώ. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί δράση όσον αφορά την ικανότητα υπεραλίευσης, γιατί θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένα δίκαιο σύστημα μεταξύ των χωρών μελών. Επίσης είναι ιδιαίτερο σημαντικό για την Πορτογαλική Βουλή να παίξει ένα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε εδώ τις δικές μας απόψεις με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε κύριε Τώρα εκ μέρους της Σλοβενίας έχουμε δύο εκπροσώπους. Καταρχήν, για την κοινοβουλευτική συνέλευση θα δώσω το λόγο, θα δώσω το λόγο στην κυρία ε, Πρέκαν. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω την Επίτροπο και τους συναδέλφους. Στη Σλοβενία υποστηρίζουμε τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και τις θέσεις που παρουσιάζονται στην Πράσινη Βίβλο. Να υπενθυμίσουμε εδώ βέβαια ότι οι προσπάθειες για να βελτιώσουμε την παρούσα κοινή πολιτική μας δείχνουν ότι για την ε, περίοδο μέχρι το 2013 έχουμε τοποθετηθεί λανθασμένα στα όσα έχουμε αποφασίσει. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια εκβάθρον μεταρρύθμιση ε, της κοινή ελευτικής πολιτικής ώστε για το χρονικό διάστημα 2014-2020 να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δύο-τρία υψίστη σημασία μέτρα πέραν των μέτρων για την υδατοκαλλιέργεια. Δηλαδή, σταδιακά μεν, αλλά με συνεκτικό τρόπο να μειωθεί η αλευτική ικανότητα, η αλευτική προσπάθεια, καταργώντας με οριστικό τρόπο συγκεκριμένες δραστηριότητες ή μετατρέποντας ε, συγκεκριμένες αλλιευτικές ε, τεχνικές με συγκεκριμένη τεχνολογία έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και τις επιστημονικές δυνατότητες που έχει μια χώρα. Για να μην υπάγεται η επιστήμη στα οικονομικά συμφέροντα. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι αλληλείς είναι άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να επιβιώνουν με τα όσα αλλιεύουν και επομένως ε, θα πρέπει να υπάρχουν κοινοτικές πολιτικές και είναι και η υποχρέωσή μας να τους βοηθήσουμε να μετατρέψουν την αλία τους. Όσον αφορά τώρα το, επιτρεπόμενο, το μέγιστο επιτρεπόμενο ελίευμα, θα πρέπει αυτό να γίνεται ανά και να λαμβάνεται υπόψη και το θέμα των νεαρών ψαριών και να μην γίνεται κάθε χρόνο ε, αναδιάθρωση για κάθε συγκεκριμένο είδος ψαριού. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα εναλλασσόμενο το οποίο να πηγαίνει εκ ε, για κάθε χρονιά. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω και να υπενθυμίσω την πάγια πρακτική της Ιταλίας, η οποία πριν από 25 χρόνια απαγόρευσε στους αλληλείς ε, την αλληλή αγώνου και μικρών ψαριών και σε εκείνο το διάστημα φυσικά είχαν δικαίωμα σε κάποια αποζημίωση. Προκειμένου βέβαια να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οι ίδιοι οι αλληλείς είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει ε, να έχουν και λόγο σε ανάλογες αποφάσεις. Ε, κάθε κράτο μέλος μπορεί να αναπτύξει εθνικά προγράμματα και εθνικά σχέδια επί του θέματος. Όσον αφορά τώρα στην ενημέρωση και στην εξοικείωση των Ευρωπαίων πολιτών με τη βιωσιμότητα τη αλληλευτική πολιτική, αυτό είναι ένα τρίτο βήμα το οποίο θα πρέπει να γίνει προκειμένου να υλοποιηθούν όλα όσα θέλουμε. Το ξέρω βέβαια ότι ε, καθυστέρησα, γι' αυτό θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Πέκα. Από πλευράς Ισπανίας τώρα Έχουμε εκπροσώπους και από τις δύο βουλές. Θα δώσω το λόγο στο Κογκρέσο στην κυρία Μαρία Αντώνια Τρουχέρο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Μαρία Αντώνια Τρουχέγιο, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Αλίας του Κογκρέσου των Βουλευτών. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόσκληση της Επιτροπής σας και για το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα να ακούσουμε όχι μόνο τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και την Επίτροπο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν από ένα μήνα στις αρχές Μαΐου έγινε ε, στο Βίγκο το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Αλληλείας στο οποίο όχι μόνο έγινε ανταλλαγή απόψεων για το κείμενο της διαβούλευσης το οποίο ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά εξετάστηκαν και προσανατολισμοί της διάσκεψης η οποία έγινε στην Ακορούνια και φυσικά ε, συζητήθηκαν και θέματα τα οποία είναι υψής της σημασίας και σχετίζονται άμεσα με την ε, μεταρρύθμιση, με την ε, ε, παράκτια και ε, μικρής κλίμακας αλίας, καθώς επίσης και εξωτερική διάσταση της αλίας μεταξύ άλλων. Θα πρέπει να πω εδώ ότι τόσο σε αυτή τη συνεδρίαση όπως και στη σημερινή φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από πλευρά όλων των αντιπροσωπιών ώστε στο μέλλον να έχουμε μια πιο βιώσιμη αλληλεία για την επόμενη δεκαετία αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι ερίζουν οι απόψεις όσον αφορά στους μηχανισμούς ε, που θα πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και οι επόμενοι μήνες φυσικά θα είναι πολύ σημαντική. Η κοινή αλληλευτική πολιτική και η μεταρρύθμισή τη θα είναι μία από τι πιο φιλόδοξε που έχουν γίνει μέχρι τούδε και θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι ώστε να μην υπάρχουν αμφισημίε. Μεταξύ στόχων θα πρέπει να έχουμε μία βιώσιμη αλληλεία που θα μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά τη και ένα ε, Αξιοπρεπέ εισόδημα για τους αλληλεί που δραστηριοποιούνται στι παράκτητε περιοχές. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα, ακούσαμε πολλές αντιπροσωπείες, αλλά εγώ θα σταθώ σε ελάχιστα εξ αυτών. Καταρχάς, ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με τους πολιτικούς στόχους της κοινή αλληλευτικής πολιτική. Να ορίσουμε με σαφή τρόπο του στόχου αυτού, διότι αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη μεταρρύθμισης ο καθορισμός των στόχων αυτής της μεταρρύθμισης, να έχουμε δηλαδή οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες βιώσιμες, ε, χωρίς να λέμε ότι ένας από αυτούς θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, διότι θα δημιουργηθούν δυσκολίες ε, ε, στον τρόπο εφαρμογής. Αυτό το τριπλό σημείο το οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε, διότι είναι πολύ δύσκολο, διότι ορισμένε φορέ οι οικονομικέ συνέπειε επιβαρύνουν το περιβάλλον ή αντιστρόφω. Η διαφορά που έχουμε σε σχέση με τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις κοινή αλληλευτικής πολιτικής είναι ότι έχουμε να λάβουμε υπόψη αυτούς τους στόχους, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Θα πρέπει να εστιάσουμε επίσης στο οικοσύστημα, αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό, και επειδή ακριβώς ε, θέλουμε να μπορέσουμε να εκμεταλλευόμαστε την αλληλεία με την αρχή του μέγιστου βιώσιμου εισοδήματος, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει ένα βήμα περαιτέρω. Η διαχείριση των απορρίψεων θα αποτελήσει επίση ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί στη μεταρρύθμιση ε, τη κοινή αλληλευτική πολιτική και για το οποίο υπάρχει ακόμα ευρεία συνένεση. Όσον αφορά τώρα στι ποσοστώσεις, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονό ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλα μοντέλα ε, της δραστηριότητα, δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα η αλληλευτική προσπάθεια, ε, αλλά δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση, διότι τα διάφορα είδη αλληλεία και αλλίευση είναι ε, πολύ διαφορετικά μεταξύ των. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια λύση η οποία θα είναι αποδεκτή μεν για τις μεγαλύτερες ε, αλλιευτικές επιχειρήσεις αλλά δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να πλήττονται οι παράκτιες ε, αλληλείας και οι μικρής κλίμακας αλληλείας διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική διάσταση και όχι μόνο την οικονομική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την Ισπανική Γερουσία. Ο κύριος Κολόμπερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές των διαφόρων χωρών μελών για να διατυπώσουμε τον ορισμό της κοινή μελλοντικής ελευτικής πολιτικής είναι αναγκαίο να δούμε ποια είναι η κατάσταση της αλίας καθώς και ο δρόμος που διανύσαμε να φτάσουμε εκεί. Η ιστορία της ε, κοινωνικής αλληλευτικής πολιτικής είναι ένα αποτέλεσμα της ιστορικής εξέλιξης της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και δεν μπορούμε να το δούμε έξω από αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να δούμε ότι σε αυτή τη διαδικασία υπήρξαν άλλοι πολιτικοί στόχοι που για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών υπήρξαν ιδιαίτερως σημαντικοί, πιο σημαντικοί από την εξέλιξη μιας κοινή ισορροπημένης και αποτελεσματικής αλληλευτικής πολιτικής. Αυτό ήταν το τίμημα που πλήρωσε η Ευρωπαϊκή Αλία, η οποία μέχρι στιγμής είδε τα αποτελέσματα της ε, πολιτικής αλίας όσον αφορά τη συντήρηση των πόρων και την οικονομική πρόοδο, τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδανικά. Ε, και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να ληφθούν αναγκαία πολιτικά μέτρα στη βάση επιστημονικών ερευνών για να πετύχουμε τα αποτελέσματα. Στη μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής εξετάζονται διάφορα θέματα. Έχω λίγο χρόνο στη, συζήτησή, ε, στη διάθεσή μου, και θα, αλλά θα θέσω ορισμένα από αυτά τα σημεία. να αναγνωρίσουμε εκείνους τους ε, στόλους που έχουν ε, υπερβολική αληφτική ικανότητα. Να ορίσουμε την αναγκαία ε, τις αναγκαίες, τους αναγκαίους στόχους ε, βιωσιμότητας και να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό ταμείο για τον παροπλισμό του στόλου. Όπως είπε η κυρία Τρουχίγιο, η κοινή ελευτική πολιτική θα πρέπει να διατηρήσει κοινωνικούς στόχους, οικονομικούς στόχους και οικολογικούς ταυτόχρονα. Μία στήριξη, μία ποιοτική απασχόληση σε αυτό το κλάδο προωθώντας τις ε, παράκτιες ε, περιοχές. Ανάγκη να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε στον κλάδο να εκπληρωθούν οι στόχοι της αλληλευτικής πολιτικής. Θα πρέπει να ρυθμιστούν τα μέτρα αυτοδιαχείρισης και αυτοελέγχου για τους ε, και να καταστούν πιο υπεύθυνοι οι καταναλωτές και να ελοπιθεί σωστή διάγνωση όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων εκπροσώπησης των αλλιέων αλλά και των ενώσεων καταναλωτών. Να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα ώστε αυτές οι οργανώσεις να μπορούν να ελοπίσουν τα μέτρα αυτοελέγχου θα πρέπει να θεσπιστούν ε, μέτρα δίκαιης αποζημίωσης ε, για την έγκριση αυτών ενός αποτελεσματικών μέτρων αυτοελέγχου. Τώρα, θα πρέπει να υπάρξει ένα διαφορετικό καθεστώ όσον αφορά την προστασία των παράκτιων ε, στόλων αλλία μικρή ε, κλίμακα, λαμβάνοντα υπόψη τι κοινωνιο-οικονομικέ επιπτώσει που επιτρέπει να διατηρήσουμε τον κοινωνικό ιστό και να εγγυηθούμε μια βιώσιμη αλία. Θα πρέπει να οριστεί η έννοια τη ε, αλία μικρή κλίμακα σε ολόκληρη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, να καταργηθεί το σύστημα της σχετικής σταθερότητας και ε, ε, ε, κατοχύρωση της ζώνης των 12, 12 μιλίων στα χωρικά ύδατα. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν τα ειδικά μέτρα για να μην ε, συνεχίσουν οι διαφορές μεταξύ αρχικής ε, τιμής και τελικής ε, τιμής για τα προϊόντα των, της αλίας. Θα πρέπει να θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε ο κλάδος να έχει την σημασία που του προσήκει ε, στην ε, ε, τροφική αλυσίδα. Θα πρέπει να υπάρξει μια ποιοτική αναγνώριση των προϊόντων και θα πρέπει να πιστοποιούνται τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Αλλά θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά ο χρόνος με εξαντλήθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Για να τελειώσουμε αυτό το πρώτο γύρο, ο θα πάρει το λόγο ο κύριος Λάρσον. Eh, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια αλλά και από το Ευρωκοινοβούλιο, από σφυδική πλευρά, θα ήθελα να πω ότι όλα τα μέρη συμφωνούν στο ότι θα πρέπει η μεταρρύθμιση αυτή να αποβεί επιτυχής και βεβαίω δεν θα πρέπει να αρκεστούμε σε ευχολόγια, θα πρέπει να δεσμευτούμε ούτω ώστε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί. Και βεβαίω θα πρέπει να ληφθούν κάποιε αποφάσει που ενδεχομένω είναι δυσάρεστε και βραχυπρόθεσμα είναι κάπω επώδυνε. Όταν μιλούμε τώρα για, τα, για τις κοινωνιοοικονομικές επιπτώσεις και τις ε, διαστάσεις μεταρρύθμισης, βεβαίως όλες οι πτυχές είναι σημαντικές εδώ. Αλλά όταν συζητάμε το θέμα αυτό στη Σουηδία, στην, ε, και το κάναμε στην Επιτροπή Αλίας, στην Αρμόδια Επιτροπή Αλίας, τότε ε, ε, λέγεται κατ' επανάληψη ότι η οικολογική βιωσιμότητα είναι η βασική προϋπόθεση για την κοινωνιοοικονομική επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Γιατί χωρίς αυτήν την οικολογική βιωσιμότητα δεν μπορούμε να πετύχουμε απολύτως τίποτε. Ένας ένα στήριγμα αυτής, βασικό στήριγμα αυτής της διαδικασίας είναι η λήψη αποφάσεων. Η απόφαση που επίκειται εδώ ε, στο Συμβούλιο Αλίας όταν οριστούν τα ποσοστά των αλλιευμάτων ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Χρειαζόμαστε πιο γενικές αποφάσεις, αποφάσεις για τις γενικές αρχές αυτό θα πρέπει να πράξουν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις και τα υπόλοιπα θέματα, οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις που είναι μάλλον τεχνικής φύσεως θα πρέπει να ληφθούν από την Επιτροπή ή σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, τέλος, από ε, ε, σουηδικής πλευράς θα θέλαμε να πούμε ότι η περιφερειοποίηση είναι μεγάλη σημασία. Υπάρχουν μεγάλες, τεράστιες διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και όταν θέλουμε εδώ να πετύχουμε υψηλά επίπεδα αποδοχής στη μεταρρύθμιση της ελευτικής πολιτικής θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι αλληλείς, οι ερευνητές, όλοι να συνενέσουν σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σωστός διάλογος με όλες τις πλευρές τους ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ένας ε, βασικός πυλώνας ε, σε αυτά τα προγράμματα διαχείρισης είναι η διεύρυνση των τομέων αλίας. Για παράδειγμα, η Βόρεια Θάλασσα, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση των υποθεμάτων και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για βιωσιμότητα. Έχει προηγηθεί βεβαίως ένας ε, προγραμματισμός. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν να λάβουν ε, υπεύθυνες αποφάσεις. Ε, εδώ δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν βραχυπρόθεσμες αποφάσεις, γιατί τα αποθέματα έπρεπε καταρχήν να ανασυσταθούν. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε τον πρώτο γύρο και η ναι. Επίτροπο ζήτησε να παρέμβει διότι θα πρέπει να φύγει. Υπάρχουν βέβαια εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής που θα μπορούσαν να παρέμβουν ε, στη συνέχεια. Να δώσω το λόγο στην Επίτροπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά τους. Ήταν μεγάλη χαρά να ακούσω από όλου εσά ε, τόσα πολλά στοιχεία και θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου να συμπεριλάβουμε την άποψη όλων. Θα ήθελα να κατανοήσετε ότι υπάρχουν κάποια θέματα για τα οποία μπορούν να γίνουν μεν πάρα πολύ καλέ συζητήσει. υπάρχουν κάποια θέματα όμω που είναι εκτό πεδίου φερμαϊκή τη μεταρρύθμισης της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι δεν μπορώ να έχω άποψη για θέματα τα οποία βρίσκονται στις συνθήκες όλοι πρέπει να σεβόμαστε τις συνθήκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εναντίον των συνθήκων, επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να σταθώ σε ευαίσθητα θέματα τα οποία είναι απόρρια μακροσκελού συζητήσεων μεταξύ κρατών μελών και αντικατοπτρίζονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις συνθήκες. Θα πρέπει να παραμείνει σχετική σταθερότητα, θα πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε την αλλαγή αυτού του θέματος αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να παραμείνει αυτό το οποίο έχουμε επιτύχει για την πρόσβαση στα χωρικά ιδίωτα υπάρχει μια κοινή αλληλευτική πολιτική. Δεν μπορούμε να επισχωρήσουμε τώρα και να επανεθνικοποιήσουμε τις αλληλευτικές μας πολιτικές. Ακόμα και αν ήθελα εγώ να το κάνω, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να το κάνω. Θα ήθελα να είμαι πολύ ειλικρινής και πολύ ανοιχτή μαζί σας. Σας παρακαλώ λοιπόν να εστιάσετε σε πράγματα, σε στοιχεία τα οποία μπορούν να αλλάξουν, μπορούμε να τα συζητήσουμε και μπορούμε να τα αποφασίσουμε από κοινού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα τώρα να σας ευχαριστήσω όλους, διότι αν κατάλαβα καλά και νομίζω ότι ε, καλά κατάλαβα, υπάρχει συμφωνία για τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους αναφέρθηκαν στην προσπάθειά μας. Υπάρχει προσπάθεια, γίνεται προσπάθεια στην Πράσινη Βίβλο και στις αποφάσεις μας να συμφιλιώσουμε όλες τις πτυχές της πολιτικής μας. Αναφέρουμε στη βιωσιμότητα, στην κοινωνική διάσταση και στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου μας. Θα πρέπει να παραμείνουμε στην προσπάθειά μας και να συνδυάσουμε αυτές τις τρεις διαστάσεις. Είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι για παράδειγμα μόνο η μία διάσταση, η βιωσιμότητα, η κοινωνική διάσταση, η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να είναι προτεραιότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Αλλά αν έχουμε μία η οποία κυριαρχεί των άλλων δεν θα έχουμε μεταρρύθμιση ή θα έχουμε μία μεταρρύθμιση με πολύ ε, περιορισμένα αποτελέσματα και εμείς θέλουμε μία μεταρρύθμιση με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, Άκουσα στοιχεία για την περιφερειοποίηση. Υπάρχουν πολλές προτάσεις ε, επί του θέματος και θα ήθελα να τις περιλάβω τις πολιτικές μας. Άκουσα πολλά στοιχεία για την ανάγκη να ενισχυθούν οι οργανώσεις παραγωγών και η ευθύνη του κλάδου. Συμφωνώ τους μαζί σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βρούμε λύσεις για το θέμα αυτό. Και επίσης υπάρχει ευρεία συμφωνία για την ανάγκη παρέμβασης στην αλυσίδα μεταξύ αλληλείας και την τελική κατανάλωση του προϊόντος στην αγορά. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα εδώ υπάρχει επιπρόσθετο όφελος, ε, προστιθέμενη αξία, πολλοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται και αποφελούνται από αυτή την αλυσίδα και ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλά ε, προβλήματα, ε, ψάρια τα οποία είναι σε καθεστώς ποσοστώσεων, τα οποία δεν καταναλώνονται ως αλλιεύματα και θα πρέπει να λυθούν πολλά προβλήματα εδώ. Με χαροποιεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επιφυλάξεις για ειδική μεταχείριση για τη μικρή κλίμακα σαλίας, θα πρέπει να δούμε βέβαια πώς την ορίζουμε την μικρή, μικρής κλίμακα αλία. Ε, α, καταλαβαίνω έχουμε διάφορες εναλλακτικέ λύσεις εδώ και θα πρέπει να καθορίσουμε απλούς κανόνες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε όλοι να κατανοούν τι θέλουμε να επιτύχουμε. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την υδατοκαλλιέργεια, συμφωνώ μαζί σας. Εάν εισάγονται τόσα πολλά ψάρια από παντού και εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την αναποραγωγή των δικών μας αποθεμάτων, πρέπει να δοθεί μια διέξοδος για τους ελλείς μας. Και νομίζω ότι οι επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου θα μπορέσει να βοηθήσει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να έχουμε πολλά προϊόντα που μπορούν να υποκαταστήσουν αυτά τα οποία θερούμε από τους άλλους κλάδους. Μια τελευταία παρατήρηση τώρα για τα ITR. Ξέρω ότι το θέμα είναι διαφιλονικούμενο αυτό που θα ήθελα να πω εδώ είναι ότι τα αλλιευτικά αποθέματα για μένα είναι δημόσιο αγαθό. Αυτό σας είπα. Γι' αυτό ακριβώς δεν ε, συζητάμε καν το να εκχωρήσουμε τα λευτικά αποθέματα σε κάποιον. Απλώς μιλάμε για δικαιώματα πρόσβασης, δικαιώματα χρήστη. Θα δώσουμε δικαιώματα σε ανθρώπους που ήδη διαθέτουν αλλιευτικά σκάφη, που σχετίζονται με τον αλλιευτικό τομέα. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και φυσικά θα το συζητήσουμε για το πώς θα υλοποιηθεί. Θέλουμε να δώσουμε δικαιώματα χρήσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 10 χρόνια, 15 χρόνια και κατόπιν, εάν αυτά τα δικαιώματα χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο, τότε θα τους ανανεωθούν. Αλλιώς ε, τα δικαιώματα αυτά θα ε, πάνε και πάλι στο κράτος. Δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση όπως άκουσα εδώ των αλληλευτικών αποθεμάτων. Συμφωνώ μαζί σας ότι τα αλληλευτικά αποθέματα είναι δημόσιο αγαθό. Γι' αυτό ακριβώς ε, μιλάμε για δικαιώματα χρήση. Φυσικά βέβαια η συζήτηση θα μπορούσε να συνεχιστεί στο δινεκές, ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις. Αυτό όμως που θα ήθελα να κατανοήσετε όλοι, θα ήθελα να το επαναλάβω για να είναι σαφές, δεν υπάρχουν κονδύλια για παροπλισμό σκαφών. Ούχαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Και επομένω να πω ότι εάν υπήρχαν χρήματα, να τα δώσουμε. Το έχω συζητήσει με τα κράτη-μέλη και ομολογώ σε εσά ότι δεν μπορώ να βρω κανέναν Υπουργό Οικονομικών από κανένα κράτος μέλος που να είναι διατεθειμένος να δώσει χρήματα για την εθνική συνεισφορά. Τι θα κάνουμε λοιπόν με τους αλληλείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε χρήματα για παροπλισμό. Εάν δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να πουλήσουν τα λεφτικά τους δικαιώματα, τι θα κάνουν. Δεν μπορούμε να τους ταξιοδοτήσουμε πρώιμα, διότι κανένας υπουργό οικονομικών αυτή τη στιγμή δεν θα συμφωνούσε σε πρόορη συνταξιοδότηση. Τι θα κάνουμε λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα να είστε λίγο ρεαλιστές όλοι. Να σκέφτεστε με πραγματικούς όρου, για το τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για τους αλληλεί, για την, υπερβολική για την υπεραλίευση, εάν δεν υπάρχει άλλη λύση. Και θα ήθελα εδώ να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Οι λύσεις που έχουμε είναι τρεις. Παροπλισμό, πρόορη ταξιοδότηση ή τα ε, ITR. Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση. Αν έχετε κάποια άλλη λύση, εγώ εδώ είμαι. Δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω περισσότερο. Έπρεπε να φύγω στις 4.30 και ήδη έχω καθυστερήσει. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας. Αν έχετε κάποια πρόταση να μου κάνετε, στείλτε μου ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προσπαθήστε να βρείτε κάποιον άλλον τρόπο. Αλλά προ το παρόν και έχω εξετάσει όλη τη διαδικασία διαβούλευση, δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη λύση η οποία να προσφέρει ταυτόχρονα βιωσιμότητα, μέγιστο επιτρεπόμενο κέρδο και κοινωνική συνοχή. Δεν μπορώ να βρω άλλο τρόπο. Γνωρίζω πολύ καλά ποιε είναι οι ανησυχίε σα, γι' αυτό ακριβώ αποσύρθηκε η πρόταση του προηγούμενου επιτρόπου τα ITR να είναι μεταβιβάσιμα σε όλη την Ευρώπη. Εγώ αναφέρομαι μόνο στα εθνικά συστήματα, ακριβώς λόγω τη σχετική σταθερότητα αναφέρομαι στην προστασία των στόλων της μικρής κλίμακας Γι' αυτό ακριβώς και δεν θα έχουμε μεταβήμαση δικαιωμάτων από μικρά σε μεγαλύτερα σκάφη, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το εθνικό σύστημα ETR από τις προοπτικές μας. Εάν βέβαια μείνετε στις θέσεις σας, θα το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και στο επανειδήν. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτός ο πρώτος γύρος. Και στο δεύτερο γύρο θα, θα υπάρξουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εν πάση περιπτώσει που αφιερώσετε το χρόνο στους Ευρωπαίους βουλευτές και ιδιαίτερα στους βουλευτές από, από τις χώρες μέλη, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. no, sí, sí, sí, sí. sí. A ver, a ver, silencio de los diputados europeos. Bueno, a ver. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε το κατάλογο για το δεύτερο γύρο όπου θα παρέμβουν οι ευρωβουλευτές. Έχουμε δέκα μέλη από, τις διάφορες, από τα διάφορα εθνικά κοινοβούλια και από το Ευρωκοινοβούλιο έχουμε 7 μέλη. Θα πάρουμε έναν έναν έναν. Λοιπόν, ε, καταρχήν, εκ μέρους της Βουλγαρίας, στον κύριο Πένκο Ατάνασοφ, Αθανάσοφ. Λοιπόν, έχουμε τρία λεπτά ομιλίες, γιατί στις 6.30 ακριβώς θα πρέπει να τελειώσουμε για δύο λόγους. Γιατί έχουμε ένα κοκτέιλ για τους προσκεκλημένους μας, όπου θα μπορέσετε βεβαίως να κάνετε επαφή με τους ε, εθνικούς βουλευτές και γιατί οι διερμηνείς θα πρέπει στις 6.30 να τελειώσουν και ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η εργασία τους. Ε, πόσο δύσκολο είναι να δουλέψουμε με μία γλώσσα. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε χρόνο σε όλους τους ομιλητές. Γι' αυτό να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας. Ο κύριος ε, Αθανάσοφ από τη Βουλγαρία. Για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Μετά την παρουσίασή μου μάλιστα πρέπει και να φύγω. Αλλά θα ήθελα να πω ότι μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα μερικά από αυτά που άκουσα. Πρώτον, μια νέα διαχείριση της αλληλείας με μέγιστη λήψη υπόψη εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Θεωρούμε ότι πρέπει η νέα πολιτική να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά να λαμβάνει υπόψη της και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Έτσι ώστε να δημιουργηθούν κριτήρια που να ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να προσαρμοστούν οι βασικές αρχές, μακροπρόθεσμοι στο σε πανενωσιακό επίπεδο με τις περιφερειακές πραγματικότητες για να μπορούν οι περιφέρειες να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν από μόνες τους τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν για να επιτευχθούν οι μακροχρόνιοι στόχοι τους δεύτερον. Η βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προς στιγμή είναι οι μόνες δύο χώρες μέλη με ακτές στη Μαύρη Θάλασσα τα αλλιευτικά αποθέματα εκεί δεν είναι γνωστά με απολύτως ακριβή τρόπο και πρέπει να έχουμε καλύτερα στοιχεία. Είμαστε βεβαίως υπέρ της αύξησης και της βελτίωσης των υδατοκαλλιεργειών διότι αυτό θα ήταν πολύ καλό υποκατάστατο για τα, τις ελλείψεις της αλίας μας. Είναι λοιπόν θέμα και διαρθρωτικό και θέμα χρηματοδότησης. Εμείς στη Βουλγαρία θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η δημόσια επιχορήγηση και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού διότι υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες που δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε χωρίς δημόσια χρηματοδότηση παραδείγματος χάρη για την υποκατάσταση του στολίσκου Επόμενο θέμα, η διαχείριση της παράκτιας αλίας, πράγμα το οποίο έχει μερικές πολιτιστικές ή και πολιτισμικές ακόμη πτυχές και αυτό σημαίνει ότι και εδώ πρέπει να καθοριστούν επίσης κριτήρια και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να διατηρηθούν τα αποθέματα, να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον και να επιτευχθεί τοπική οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επιτραπούν πλοιάρια μήκους μέχρι και 12 μέτρων που να αλλιεύουν μέσα στην, στα 12 μίλια. Η κυρία Ανδρές Παρέα, ευχαριστώ. Να σας συγχαρώ κυρία Πρόεδρε για αυτή την πρωτοβουλία, διότι έτσι μπορούμε να γνωριστούμε οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές ε, από τα διάφορα κράτη-μέλη θεωρώ ότι βρισκόμαστε ενώπιον μια σημαντική μεταρρύθμιση τη κοινή μία μεταρύθμιση την πολιτική. Ε, μια μεταρρύθμιση την οποία επεξεργαστήκαμε. Είχαμε μια πολύ καλή έκθεση. Μια έκθεση που αναφέρεται σε δικαιώματα και σε εγγυήσει. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα ώστε η μεταρρύθμιση να είναι συνεκτική και να είναι και μακροπρόθεσμη. Αλλαγή στη διαχείριση, πολύ σημαντικά τα τάκια ποσοστώσεις και οι απορρίψει και να αλλάξει ο τρόπο διαχείρισή του. Η συμπλήρωση της αγοράς ε, που σημαίνει ότι οι κοινέ οργανώσεις ε, αγοράς των αλλιών θα είναι πολύ σημαντικά. Ε, τώρα τα ατομικά δικαιώματα αλλιάς τα οποία μπορούν να μεταβιβάζονται, τα ITRs, είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται ε, συζήτηση για τη μικρή κλίμακα αλεία θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κερδοσκοπία. Η Κομισιόν ήταν πολύ συγκεκριμένη. Είναι ένα μέσο εμπορία κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουν, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που γινόταν ήταν να παίρνει κάποιο την άδεια από τη μία και να την πουλά από την άλλη. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέτρο αυτό, μπορούμε να το εξαντλήσουμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όρια και θα πρέπει να το μελετήσουμε ως δυνητική λύση. Τώρα, οι διεθνεί συμφωνίε τι οποίε υποψιαζόμαστε συνεχώ, κυρίω η Διεθνή Συμφωνία Αλία, διότι για τα ε, υπόλοιπα, ε, θέματα δεν θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι τόσο ύποπτα, θα πρέπει να βρούμε την ηθική αξία αυτών των ε, συμφωνιών, διότι βοηθούν στην ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό των χωρών αυτών. Η κοινή αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να αποτελεί λύση κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική είναι σαφές ότι στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε θα πρέπει να είμαστε αυτάρκεις και να βλέπουμε προς το μέλλον για να έχουμε μία λύση ε, για τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να θέσουμε θέματα τα οποία όχι μόνο να μας αφορούν προσωπικά αλλά και να απευθύνονται στο σήμερα αλλά να δούμε στο μέλλον, στο αύριο. Εγώ ευχαριστώ κύριε Άντρες Μπαρέα και τώρα εκ μέρους της Γαλλίας η κυρία Λέλοπ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω τρία ερωτήματα να θέσω στην κυρία Επίτροπο. Η Γαλλία είναι πολύ κριτική όσον αφορά την υπεραλίευση. Ε, τι γίνεται με τις ποσοστώσεις η Βρετάνη έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες με δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις. Πώ η περιφερειοποίηση, όπω ανέφερε προηγουμένως η κυρία Επίτροπο, μπορεί να, γίνει, να καταστεί πιο δίκες ε, να καταστήσει πιο δίκαιες αυτές τις ε, προσπάθειες. Η ε, κοινή ελευτική πολιτική ίσως θα έπρεπε να παράχει τη δυνατότητα μιας πιστοποίησης των απορρίψεων για να μην ε, υπάρχει και αύξηση των ε, εισαγωγών των ψαριών. Και τρίτον, κυρία Επίτροπη, αναφέρετε συχνά τη μοίρα των ε, παράκτιων κοινοτήτων και βλέπω μια απουσία ανθρώπινης διάστασης στην πολιτική μια βιώσιμη πολιτική δεν μπορεί να γνωρίσει αυτή την ανθρωπιστική διάσταση και την κοινωνική πτυχή. Πώς ε, θέλετε να τη συμπεριλάβετε στην ε, δική σας πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λελόκ. Στη συνέχεια ο, ο κύριος Κάντεκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση ήταν αναγκαία γιατί επιτρέπει στους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια να μπορούν να έχουν μια ανταλλαγή απόψε με εμά και να έχουν ένα σημαντικό επίπεδο πληροφόρησης. Έχουμε περισμένο χρόνο ομιλίας, γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω στη συνάδελφα από τη Βρετάνη γιατί ανέφερε το ζήτημα των εισαγωγών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μας διαφεύγει γιατί η Ευρώπη εισάγει 60% της κατανάλωσης, κάτι που είναι τεράστιο. Και συνεπώς ε, θεωρώ αν τα θέλουμε να διαφυλάξουμε ή να διατηρήσουμε τη δική μας αλία είναι αναγκαίο να εφαρμόσουμε τους ίδιους ε, περιορισμούς στις αγωγές που επιβάλλουμε στους δικούς μας αλείς, τουλάχιστον γιατί είναι θύματα θέμη του ανταγωνισμού στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε μια περιβαλλοντική και υγειονομική χνηλασιμότητα για όλα αυτά τα προϊόντα. Για παράδειγμα στα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας από την από Ανατολή που κατακλείζουν τα ράφια των καταστημάτων μας και θα πρέπει να τα ε, επισημάνουμε ως ευαίσθητα προϊόντα, αυτά τα προϊόντα της ηχθειοκαλλιέργειας για να διατηρήσουμε ένα λογικό επίπεδο επίπεδο των ε, τελωνιακών ε, δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι αντικείμενο μια έκθεση που θα παρουσιάσω στην Επιτροπή στις 22 Ιουνίου, αγαπητοί συνάδελφοι, και ελπίζω στο Κοινοβούλιο στις αρχές Ιουλίου και ελπίζω ότι ε, θεωρώ ότι αυτό αφορά την επιβίωση των αλλιών μας, γιατί αν δεν ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα των εισαγωγών, μπορούμε να κάνουμε σκέψεις ε, περί δικαιοσύνης ή περί τεχνικών μέτρων, αλλά αν ρυθμίσουμε το ζήτημα των εισαγωγών, σε 10-15 χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε ένας Ευρωπαίος αλλιέας. Κατά τα άλλα είμαι σύμφωνος με τα όσα υπόθηκαν εδώ και συμμερίζομαι, επειδή θεωρώ ότι η απάντηση της Επιτρόπου όσον αφορά τα ατομικά μεταβάσιμα δικαιώματα, όχι στο επίπεδο της Ευρώπης, αλλά στο επίπεδο της κάθε χώρας, μπορεί να είναι μια αποδεκτή απόκριση ή, εν πάση περιπτώσει, μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Ιδού, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Με χαροποιεί αυτό, κύριε Κάντεκ. Είπα σε εθνικό επίπεδο. Είπα ότι προχωρούμε προς κατάσταση που είναι θετικό. Το λέω για να γνωρίζουν και οι βουλευτές ότι και εμείς εδώ έχουμε τις διαφωνίε μας, αλλά παρά αυτά καταφέρνουμε να προχωράμε και να επιτυχάνουμε συμβιβασμού. Είπα σε εθνικό επίπεδο, ε, να λαμβάνει ο κύριο Κάντε. Σας άκουσα κύριε Κάντε, γι' αυτό λέω ότι προχωράμε. Σε εθνικό επίπεδο ίσως να μπορέσουμε να επιτύχουμε και άλλα πράγματα. Χαίρομαι πάντα που σας ακούω. Ό,τι ακούμε μας κάνει πάντα να σκεφτούμε αλλά πολεμάμε για μια λευτική πολιτική που μπορεί να έχει κάποιο μέλλον. Από πλευράς Γαλλίας και πάλι πηγαίνουμε αλφαβητική σειρά ε, στα κράτη-μέλη για τους ευρωβουλευτές ε, με τη σειρά ετήσεως. Από Γαλλία ο κύριος Λεκόμ λοιπόν. Συγγνώμη, Λεκού. Εγώ δεν κατάλαβα καλά το όνομα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να εκφράσω δική μου άποψη σχέση με τη Μεσόγειο, ξεκινώντας από τη Μεσόγειο γιατί είμαι βουλευτής της Μεσογείου. Θα ήθελα να σας πω ότι θεωρούμε ότι ο Αλίας είναι ο καλύτερος παρατηρητής των θαλασσών και σήμερα ο, Αλιά, ο, ε, δεν καταλαβαίνει πολύ καλά αυτό τον κανονισμό που θεωρεί ότι έχει εκπονηθεί στη βάση των χαρακτηριστικών της Βόρειας Θάλασσας, του Ατλαντικού ή της ε, Βαλτικής. Γι' αυτό λοιπόν θα ήμουν υπέρ μιας περιφερειοποίησης πολύ ξεκάθαρα γιατί η κατάσταση απαιτεί να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα της ε, θάλασσας και η πραγματικότητα της Μεσογείου θάλασσας διαφέρει από αυτή των άλλων θαλασσών. Και αν δεν το κάνουμε δεν θα υπάρχει επαρκής κατανόηση. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν στο πλαίσιο της εκπόνησης του κανονισμού της, ε, των ε, αλλιέων της Μεσογείου όπου έχουν απαγορευτεί παραδοσιακές μέθοδοι αλίας Euh, μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην Ιαπωνική, στον Ειρηνικό για την αλία των ε, δελφινιών. Ενώ στο Μεσόγειο έχουν υπάρξει απαγορεύσεις παραδοσιακής αλίας όπου το σύστημα ε, πανάρχιας ε, οργάνωσης ήταν ένα σύστημα που λειτουργούσε πολύ καλά όπου οι ελείς μπορούσαν να αυτορυθμίζονται και εφόσον ε, ο ψαράς είναι ένας καλός παρατηρητής, είναι κάποιος ο οποίος θα μεταδώσει στο γιο του την ικανότητα να, γίνεται, να είναι και αυτός ένας καλός ψαράς. Τώρα, όσον αφορά τον ανταγωνισμό των χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες, γιατί πράγματι οι κανόνες δεν είναι οι ίδιοι. Θα πρέπει λοιπόν εμείς οι Ευρωπαίοι να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί οι δικοί μας αλείς δεν ε, κατανοούν ε, πάντοτε τα πράγματα. Τέλος, ε, το θέμα του, του παραπλησμού των πλοίων. Πόσο αλλιές ε, μπορεί να καταλάβει ότι πριν από μερικά χρόνια η Ευρώπη χρηματοδοτούσε τα λεφτικά σκάφη, ενώ σήμερα δεν το κάνει. Για παράδειγμα, τον κόκκινο τόνο. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ε, πώς να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που κάποια στιγμή παρατρέθηκαν να χρησιμοποιήσουν μια συγκεκριμένη μέθοδο αλίας. Τώρα, όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, μου φαίνεται ότι είναι μια λύση, αλλά θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα ε, την εντατοκαλλιέρεια στις παράκτιες ε, περιοχές, ε, τα στρίδια συγκεκριμένα, όπου υπάρχουν ειδικά προβλήματα. Και θα ήθελα να τονίσω το θέμα της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ αλλαίων και επιστημονικών κύκλων. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Ρόμπαρτσικ από Πολωνία. E, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Αλέν αν έχει ήδη πέσει η Βαστήλη ή... και γι' αυτό μιλάτε ακόμη για το ITQ. Α, όχι, εντάξει, καλά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου της Εσθονίας και του συστήνω να διαβάσει την ιστορία της Ισλανδίας η οποία κάποια στιγμή εφάρμοσε το ITQ με αποτέλεσμα την κυριολεκτική καταστροφή της βιοτεχνικής της αλληλείας. Εξάλλου και ο κύριος Πόηρο από το Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης επιβεβαίωσε την πραγματικότητα αυτή. Είναι πολύ επικίνδυνο για την βιοτεχνική αλληλεία να εφαρμόζεται το σύστημα των ITQ. Είχαμε οργανώσει μια αποστολή για το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε καθώς και τη Γραμματεία για την εξαιρετική οργάνωση εκείνης της αποστολής Τώρα όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που μας είπαν οι αλληλείς κατά την αποστολή εκείνη που παραπονούνταν γιατί οι μεγάλες εταιρείες μεταποίησης των αλληλευτικών προϊόντων τελικά κατέστρεφαν τη δραστηριότητά τους ενώ θέλουν να συνεχιστεί προφανώς είχε καταστρεφικές επιπτώσεις και επί αυτών η εφαρμογή του συστήματος των ITQ. Σε προηγούμενη συναντρίαση είχαμε πει ότι το Πολωνικό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα την άδεια και από τη Βουλή και από τη Γερουσία την οποία εκπροσωπούν, οι οποίες εκπροσωπούνται σήμερα εδώ να δίνει την άδεια σε ψαράδες της Βαλτικής να αλλιεύουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της κοινοτικής αλληλείας. Σας ζητώ λοιπόν να σταματήσουν πια αυτοί οι πειραματισμοί. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα το οποίο έθεσα και εγώ την προηγούμενη φορά. Εσείς δεν το δεχτήκατε, αλλά ε, είναι ένα παράδειγμα που και μου είπατε ότι είναι παράδειγμα το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Τέλος πάντων. Ακούσαμε τον κύριο Βέτσεκ και τώρα να ακούσουμε έναν από τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, η κυρία Κορνίλια Μπέμ από τον Bundestag. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ρητά την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της Πράσινης Βίβλου ακριβώς εν ώψη της δυσχερούς ε, κατάστασης των ε, εχθιαπεθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ εκπροσωπώ τους πράσινους στο, στη Γερμανική Βουλή, στο Bundestag και θα ήθελα να τοποθετηθώ επί ορισμένων σημείων της πράσινης βίβλου. Θεωρούμε ότι το σύνολο των αλευμάτων, των επιτροπών αλευμάτων θα πρέπει να ορίζονται στη βάση επιστημονικών δεδομένων και δεν θα πρέπει να είναι πλέον αντικείμενο ε, διαπραγμάτευσης μεταξύ ελευτικών ε, ε, κύκλων και ομάδων συμφερόντων. Ε, όσον αφορά τα παρεπίμπτοντα αλλιεύματα, όλα τα αλλιεύματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις ε, και να υπολογίζονται. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο αποφυγής των παρεπιπτόντων αλλιευμάτων και της εισαγωγής κάποιων καινοτομιών. Έστω και για να είμαστε ρεαλιστικοί, ένα ορισμένο ποσοστό των αλλιευμάτων δεν είναι δυνατόν να αποφευθεί εντελώ. Είναι σημαντικό να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων ειδών γιατί ε, ε, θα πρέπει να αυξηθούν τα ποσοστά επιβίωσης ε, και θα πρέπει να αποφευθεί η εξάντληση των αποθεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το σύστημα των ΤΑΚ και του, ελάχιστου, του ορισμού ελάχιστου μεγέθους των αλευόμενων ηχθείων ε, μέχρι στιγμής ε, δεν είχε πολλές επιτυχίες. Απειλούνται τα αποθέματα είτε επειδή οι Υπουργοί Αλίας αυξάνουν αυτά τα ποστά επιτρεπόμενων αλλιευμάτων, είτε επειδή υπάρχει ε, παράνομη αλεία. Τώρα, όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση, χαίρομαι που η Επίτροπος μιλάει για δικαιώματα χρήσης και όχι πλέον για ιδιωτικοποίηση. Χαίρομαι που μιλάει για την αλεία σε ένα δημόσιο αγαθό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε ότι να μην υπάρχουν φαινόμενα συγκέντρωση υπέρ ορισμένων ισχυρών ε, κεφαλαίων. Η, τα αποθέματα των ηχθείων θα πρέπει πράγματι να θεωρηθούν ε, δημόσιο αγαθό και στη θέση ιδιωτικοποίηση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδέει την ετήσια διανομή των ελευτικών δικαιωμάτων ε, με ένα σύστημα επιβολής ε, τελών και με τον τρόπο αυτό θα δοθεί ένα κίνητρο για περιορισμό των ελευμάτων θα πρέπει να όλα τα μέτρα πρώτης τις να έχουν ένα οικολογικό προσανατολισμό, για παράδειγμα απαλλαγή από φόρους ε, σε παροπλιζόμενα για παροπλιζόμενα σκάφη. Θα πρέπει να βελτιωποιήσουμε τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελλοντικά να μπορούμε να ελέγχουμε τις ε, αλληλευτικές ε, συμφωνίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Καντέκ. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να παρέμβω εντάχει για να διευκρινιστεί κάτι. Εγώ είμαι κατηγορικά αντίθετος στο εξή. Ο φίλο ε, Ρόμπερτ έφυγε, αλλά η Βασιλή δεν έχει πέσει. Και δεν έχω την άποψη να αλλάζω γνώμη σαν τα αποκάμισα. Θα ήθελα να πω ότι η πρόταση τη Επιτρόπου είναι μια προόδο τη Επιτροπή προ την εγκατάλειψη τη αρχή αυτή. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως και το επαναβεβαιώνω κυρία Επίτροπε. Δεν θα απαντήσω τώρα στη δεύτερη παρέμβαση γιατί δεν θέλω να ξαναπαρέμβετε. Στη συνέχεια, μετά θα μιλήσουμε όμως, μην ανησυχείτε, δεν σας ξεχνάω. Στη συνέχεια λοιπόν, τον εκπρόσωπο της Λετωνίας, Μαρτίνς Ρόσεκ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ λίγο στη διαδικασία. Διότι στον προηγούμενο γύρο κάτι έγινε και το ΕΛ το ξεχάσατε. Η μεταρρύθμιση της κοινής ελευτικής πολιτικής είναι πάρα πολύ σημαντική Πρέπει να δώσουμε επίσης τη δέουσα προσοχή στη μείωση του διοικητικού άχθους. Ενώ ταυτόχρονα θα προσπαθούμε να έχουμε ένα απλό και διάφανο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, η αρχή της περιφερειοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η συζήτηση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τις προσδώσουν περισσότερη ουσία. Θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο οι χώρες που συμμετέχουν στην αλληλεία στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό θα διευκολύνει και το ρόλο των εθνικών εμπειρογνωμόνων. Η βιωσιμότητα είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της αλίας, αλλά οποιασδήποτε δράσεις περιοριστικές θα πρέπει να συνοδεύονται και από μέτρα αποζημίωσης για να μπορέσουμε να διασφαλίζουμε το εισόδημα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Λατανία είχε θαλάσσια σύνορα άνω των 150 χιλιόμετρων. Επομένως, πολλές περιοχές εξαρτώνται από την παράκτια Η βιωσιμότητα της ε, παράκτιας κοινωνίας θα πρέπει να προκύπτει από τη δυνατότητα που τους δίνουμε να προγραμματίσουν το μέλλον τους τα χωρικά είδητα των 12 μιλίων θα πρέπει να διατηρηθούν ε, και να επιτρέπεται να αλλιεύει μόνο ο εθνικός στόλος, εκτός και αν υπάρχει ξεχωριστή διμερή συμφωνία μεταξύ χωρών. Επίσης θα πρέπει να παραμείνει η αρχή της σχετικής σταθερότητας, βάσει της οποίας ε, τα αλλιευτικά δικαιώματα κατανέμονται βάσει ιστορικών παραγόντων. Γεγονός που σημαίνει ότι η υπεραλίευση θα μειωθεί γιατί δεν θα μπορούμε να έχουμε παραλήψεις σε ξεχωριστές ε, περιοχές. Τώρα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ε, συνδυάσει το στόλο τους ανάλογα προς την ε, διασυνθημότητα των αλλιευτικών αποθυμάτων μπορούν να αλλιεύσουν με καλύτερες προϋποθέσεις ε, σε αντιπαράθεση φυσικά με τις χώρες που δεν έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο και δεν έχουν ε, εξισορροπήσει το, στόχο τους, το στόλο τους με την αλλιευτική τους δυνατότητα. Όσον αφορά τώρα την αλίευση σε ύδατα τα οποία είναι εκτός ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας, θα πρέπει να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρακτική κάποια τεχνική οργάνωση ελίας θα πρέπει να υπάρχει κεντρικά και να υπάρχει μια κεντρική αλληλευτική υπηρεσία που θα κάνει τον έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει ε, αποστέλλοντας εθνικούς εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Αυτό θα ενισχύσει ε, και θα βελτιστοποιήσει τον έλεγχο ε, χρηματοοικονομικής συνδρομής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί και η υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων, διότι δεν μπορούν όλες οι χώρες να έχουν υδατοκαλλιέργεια θανάσεων υδάτων για γεωγραφικούς ή και ιστορικούς λόγους. Η επέκταση των ITQ θα πρέπει να γίνεται μόνο στα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή μεταξύ ε, αλλιέων ή μεταξύ χωρών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια, ο κύριος Φερέιρα από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τους εκπροσώπους των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαμε σήμερα είναι ότι εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες και ενστάσεις που είναι όλες ιδιαίτερως ε, σημαντικές και θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη. Όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από την Επιτροπή. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων να τους ζητήσω να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τους προσεχείς μήνες τη συζήτηση την εξέλιξη της συζήτησης, ιδιαίτερα όσον αφορά το τελευταίο ήμιση αυτού του έτους. Θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του θέματος, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, για λόγους χρονικού περιορισμού, θα θέσω μόνο το θέμα της πυραλίευσης και των ατομικά μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων. Ορισμένοι ε, αρκετοί ομιλητές αναφέρθηκαν στο ζήτημα της υπεραλίευσης λέγοντας ότι η πραγματικότητα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Νομίζω κάποιος από τη γερμανική Bundestag είπε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό στόλος, υπάρχουν εθνικοί στόλοι και η εθνική αλληλευτική στόλη τις τελευταίες δεκαετίες είχαν ε, διαφορετικές εξελίξεις όσον αφορά την υπεραλίευση σε ορισμένες ε, περιπτώσεις. Και η Επίτροπος αναφέρθηκε σε αυτό το φαινόμενο, ειδικά στο πλαίσιο της ακρόασης που είχε πριν από τον διορισμό της, πριν από την εκλογή της και αναφέρθηκε στις προσπάθειες των χωρών μελών ε, για τη μείωση της υπεραλίευσης και των συνεπειών της. Και βεβαίω ο αντίκτυπο ε, τη προσπάθεια αυτή ήταν πολύ διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Τώρα, όταν μιλούμε για την υπεραλίευση με γενικούς όρου, όπω γίνεται στην Πρασινή Βίβλο, τελικά δεν ε, αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα αυτού του φαινομένου όσον αφορά τα αποθέματα, του στόλους και τον εξοπλισμό των αληφτικών σκαφών. Ε, ε, χωρίς λοιπόν να εκτιμούμε αυτές τις διαφορετικές ε, εκφάνσεις της επεραλίευσης, ε, δεν νομίζω είναι καλός τρόπος να κινηθούμε προς τα μπρος. Τώρα, όσον αφορά τα ITR, τα ατομικά μεταβάσιμα δικαιώματα, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο πρότεινε η Επιτροπή ως θέμα υποσυζήτηση, παρουσιάζεται συνεχώς ως μοναδική λύση, χωρίς να υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί αυτά τα ITR, τα ατομικά μεταβάσιμα δικαιώματα, δεν είναι η δυνατότητα. Ο εισηγητή στην Πράσινη Βίβλο λέει ότι υπάρχει μια πλατιά συνένεση όσον αφορά τι καταθυντήριε Γραμμέ. Αυτό μεν αληθεύει αλλά από την άλλη κάθε ειδική μνήμα στην έγκριση των ατομικών μεταβάσιμων δικαιωμάτων έχει αφαιρεθεί από το σχέδιο έκθεσης, ούτως ώστε να διατηρηθεί αυτή η συμφωνία. Όσον ε, Θα μπορούσα να πω πολλά άλλα πράγματα, αλλά επιτρέψατε μου να πω κλείνοντα ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση και αυτό θα το υπομορφεί ερωτήσεως, Εάν ένα επενδυτή ή ένα εργοδότη από μια χώρα μέλο θέλει να αγοράσει δικαιώματα από μια άλλη χώρα μέλο, δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για το πώ θα δουλεύει κάτι τέτοιο. Eh, Εκ μέρου τη Ρουμανία ζήτησε το λόγο ο κύριος Μάριον Άμπραμ για τρία λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, Εκπροσωπώ την Ρουμανική Βουλή και ιδιαίτερα την Επιτροπή Γεωργίας της και την Κομιτεία της Δούλτσα, δηλαδή στο Δέλτα του Δούναβη, όπου βρίσκονται οι περισσότερες αλλιευτικές δραστηριότητες της Ρουμανίας. Έχουμε ένα πολύ λεπτομερές αλλιευτικό πρόγραμμα που το διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου και θεωρούμε ότι το σημαντικότερο στοιχείο του προγράμματος αυτού είναι το γεγονός ότι τα αποθέματα της Μαύρης Θάλασσας μειώνονται. Το αλλιευτικό αυτό πρόγραμμα, το σχέδιο δράσης, προβλέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλληλείας και των βοηθητικών υπηρεσιών και ε, έχει γίνει σε συνεργασία με τις οργανώσεις των ίδιων των αλλιέων. Τώρα για την πράσινη βίβλο. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας ως λύσης στο πρόβλημα της μείωσης των αποθεμάτων. Επίσης θέλουμε να αυξηθεί η συνεργασία με τη Βουλγαρία ως στα πλαίσια της κοινής πολιτικής και της περιφερειακής διαβούλευσης. Επίσης στοχεύουμε σε καλύτερους και σαφέστερους κανόνες για την ιχνηλεσιμότητα και τις συσκευασίες. Όλα αυτά θα θέλαμε να τα εξετάσουμε λαμβάνοντας υπόψη μας βέβαια και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και βιωσιμότητας όπως είπα διατήρησης της αλληλευτικής δραστηριότητας που είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα εκεί χωρίς να παραλείπουμε και την διατήρηση όλων των υπηρεσιών που χρειάζεται να στηριχθούν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα εξ ονόματος του Ευρωκοινοβουλίου η κυρία Λεβέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ήρθαν εδώ και είπαν τόσα ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μια απόφαση που είχε ληφθεί η ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα όπου προβλεπόταν ο σεβασμός των οικολογικών προδιαγραφών για τη θάλασσα, πράγμα που δεν πρέπει να το αγνοούμε όταν μιλάμε για την αλληλεία. Η αλληλεία δεν είναι το κυριότερο στοιχείο της θαλασσίας πολιτικής της Ένωσης, αλλά ένα από τα στοιχεία. Όσο για την πιθανή δυνατότητα ατομικής μεταβίβασης των ποσοστώσεων, θεωρώ ότι πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είδη αφορά η δυνατότητα αυτή, ποια ψάρια. Η Επίτροπος είπε ότι οι αλλιευτικοί πόροι είναι δημόσιοι πόροι. Πρέπει να το δούμε όμως αυτό, πώς θα τους διαχειριστούμε. Το δικαίωμα στην αλληλεία σχετίζεται με τη δυνατότητα του αλλιέως να αποδείξει ότι αλλιεύει βιώσιμα και προστατεύει το περιβάλλον. Όπως είπε κάποιος συνάδελφος, στη Δανία δίνεται προτεραιότητα στους αποτελεσματικότερους αλληλείς σε όσους χρησιμοποιούν λιγότερα καύσιμα κτλ. Αυτό ίσως είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να το ακολουθήσουμε όσο για τις επιχορηγήσεις για την απόσυρση ορισμέν, της ορισμένων ειδών και εδώ θεωρούμε ότι είναι κίνητρο, θα έπρεπε να είναι κίνητρο η χρησιμοποίηση ως το δυνατόν λιγότερων καυσίμων, ενώ η επιχορήγηση των καυσίμων είναι αντικίνητρο. Δεν ωφελεί ούτε τη θάλασσα ούτε κανέναν. Και είναι ενθάρρυνση για να συνεχίζεται η υπεραλίευση. Όσο για την οικολογική σήμανση των ψαριών και των νυχθείων πρέπει να πούμε ότι θέλουμε να γνωρίζουμε την προέλευση τους. Ο καταναλωτής και η καταναλώτρια το θέλουν και πρέπει ο αλιεύς να μπορεί να το δηλώσει προς τον καταναλωτή και την καταναλώτρια. Οι αλλιευτικές συμφωνίες πρέπει να υπογράφονται μόνον με χώρες που έχουν αποδείξει ότι αλλιεύουν με το σωστό τρόπο. Και συμφωνώ με αυτά που είπε η Γερμανίδα κυρία Μπρέμ. Ευχαριστώ. Τώρα εκ μέρους της Σλοβακίας ο κ. Λοβάσκη. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα μιλήσω από την άποψη της ε, Σλοβακίας όπου θεωρούμε ότι ο τομέας της ε, υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστό πυλώνα της κοινή αλληλευτικής ε, πολιτικής με ιδίους στόχους. Αυτή είναι η άποψη της ε, Σλοβακίας, γιατί είμαστε περιοτική χώρα. Έχουμε την άποψη ότι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, έχει αποδειχθεί ε, θα πρέπει να αποδειχθεί η καρκινογόνος επίδραση του μαλαχίτη ή να απορριφθεί ή επίσης, ε, και επίσης μια υπερσυγκέντρωση αυτής της ουσίας ε, σε σχέση με τη χρήση της στις ε, υδατοκαλλιέργειες. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες να ελέγχονται σε παρκή βαθμό. Επίσης είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η φυστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά ε, τις προδιαγραφές ασφαλείας των τροφίμων θα πρέπει να τηρείται. Και ε, ε, επίσης στον τομέα των, της γλυκού νερού δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ισορροπία μεταξύ διαφύλαξης κάποιων θηρευτών όπως είναι η κορμεράνη και της προστασίας των αποθεμάτων των ηχθείων ε, θα πρέπει να διατηρείται, να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της διατήρησης αυτών των δύο ε, των ε, πουλιών και των ψαριών. Ευχαριστώ από το Κοινοβούλιο κύριος Γκάλαχερ, Ιρλανδός, Ευρωβουλευτής. Καταρχάς να πω ότι πιστεύω ότι η σημερινή συνεδρία ήταν πολύ σημαντική ως ανταλλαγή απόψεων, πολύ χρήσιμη από πλευράς μου. Άκουσα και τη συνεισφορά των Ιρλανδών ε, βουλευτών που εκπροσωπούν ε, την Ιρλανδική αντιπροσωπεία και είπαν αυτά που λέω και εγώ κάθε μέρα. Δεν θα καθυστερήσω περαιτέρω τη συζήτηση, αλλά ακούγοντας και όλους ε, όσους ε, εκπροσωπούν τη χώρα του σήμερα, η περιφερειοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Επίτροπος λέει ότι δεν μπορούμε να ε, επανέλθουμε στην περιφερειοποίηση. Η περιφερειοποίηση δεν είναι αποκέντρωση, είναι κάτι το οποίο βοηθά τους πάντες είναι κάτι το οποίο θα προκύψει από όλου ε, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τη μικρή κλίμακα και επομένω θα πρέπει να του δώσουμε μια ειδική θέση στην ε, αναθεωρημένη κοινή αλληλευτική πολιτική, κυρίω στα μικρά παράκτια κράτη, διότι τα μικρά σκάφη αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το 80% των σκαφών μα είναι κάτω των 15 μέτρων και δεν έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις ε, στη διαχείριση των αποθεμάτων. Η Συμφωνία της Χάκης είναι πάρα πολύ σημαντική και ε, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αναθεωρημένη κοινή αλληλευτική πολιτική. Τα τάκ και οι τώρα. Δεν είναι τέλεια βέβαια. Και εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει όμως ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διαχείριση το, τα τάκια υποσωστώσει θα πρέπει να είναι ένας βασικός πυλώνας της ε, μεταρρυθμισμένης κοινή αλληλευτική πολιτικής. Ω προ το σύστημα των απορρίψεων και την απαγόρευσή τη, σαφώ δεν θα πρέπει να υπάρχουν απορρίψει. Αλλά όταν θέσουμε ω στόχο τι μηδενικέ απορρίψει, δεν θα τον επιτύχουμε ποτέ. Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε οι αλληλεί να γνωρίζουν ότι αν αλλιεύσουν ε, ε, αλλιεύματα τα οποία δεν θα έπρεπε, θα λάβουν μια κάποια αποζημίωση γιατί θα τα εκφορτώσουν για την υδατοκαλλιέργεια τώρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τη υδατοκαλλιέργεια και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εισάγουμε ψάρια από τρίτες χώρες, θα μπορούσαμε να το αντικαταστήσουμε αυτό με την ανάπτυξη της ιδετοκαλλιέργειας. Και φυσικά, ποιος γνωρίζει τερά τα πράγματα αυτά. Μπορεί να μην είναι επιστημονικό μεν ο τρόπο που έχουν λάβει τι γνώσει, αλλά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι οι γνώσει οι οποίε προκύπτουν από του ίδιου του αλληλεί, που είναι παραγωγή και αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν τα μάλλα σε όλες τις επιστημονικές πληροφορίες που έχουμε και αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί με κάποιο τρόπο και θα πρέπει να τους δοθεί μια νομική βάση ώστε να μπορέσουν να το επιτύχουν. Πολλοί αναφέρονται στα ατομικά μεταβιβαζόμενα δικαιώματα, τα ITRs. Εγώ είπα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προκειμένου να εισεχθούν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εγκρίνει κάθε κράτος μέλος. Και ξέρω για τη χώρα μου, για την Ιρλανδία, ότι δεν θα περάσει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε χρήματα για πρόορη ε, συνταξιοδότηση. Θα πρέπει να δούμε και τις εκθέσεις που είχαμε στο παρελθόν. Αν δεν έχουμε χρήματα θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να το επιτύχουμε. Διότι οι αλληλείς μπορούν να φύγουν στα 55 χρόνια, τους δίνεται μια δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν και να δώσουμε νέες θέσεις εργασία στους πάρα πολλούς νέους αλληλείς που θέλουν να εμπλακούν ε, στον κλάδο. Συμπερασματικά λοιπόν θεωρώ ότι ήταν μια καλή ημέρα η σημερινή και το γεγονός ότι η Επίτροπος ήταν διατεθειμένη να μας ακούσει και θέλει να συμπεριλάβει τις συνεισφορές μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια τώρα από την Ισπανία ο κύριος Γκαρσία Δίαθ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χωακίν Γκαρσία Δίεθ, εκπρόσωπος ε, συντονιστής αλίας ε, του ε, Παρτίδο Ποπολάρ. Ε, προέρχομαι από τη Γαλλικία. Με την άδεια της Προεδρίας θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι φέτος είναι το ιερό έτος ε, της Κομπεστέλα και ίσω θα μπορούσατε να ξεχάσετε τα προβλήματα της Ελίας, να έρχετε να προσκυνήσετε στη Σαντιάγο Δε και να δοκιμάσετε και υπέροχα ψάρια. Ε, σε αυτό μεταφράζεται η πρόσκλησή μου. Σήμερα το απόγευμα μιλήσαμε για τα προβλήματα του ελευτικού τομέα και αυτό ο τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικός για την περιοχή μου, για την Ισπανία εν γέννη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε από τους ε, επικεφαλείς, είμαστε η χώρα η οποία καταναλώνει περισσότερο ψάρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές περιοχές οι οποίες εξαρτώνται από την αλία και επομένω όλη αυτή η συζήτηση και μας ανησυχεί και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η... Μαρία Αντόγια Τροχέρο, συνάδελφος από, το, από τη Γερουσία, ε, επεσήμανε πόσα προβλήματα συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις του Βίγκο και στην Λακορούνια και το κόμμα μου, το Παρτίδο Ποπολάρ, ε, έχουν εκπονήσει και έχουν ε, προσφέρει στη συζήτηση έγγραφα τα οποία θα μπορούσα κάλλιστα να σας δώσω για να τα διαβάσετε αν το επιθυμείτε. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ την πρόεδρο της Επιτροπής, τη φίλη μου την Κάρμεν Φράγα για αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως επεσήμαναν εδώ πολλοί από τα μέλη, από τα Εθνικά Κοινοβούλια που είχαμε εδώ, διότι η συζήτηση αυτή δεν είναι μια συζήτηση κυβερνήσεων, είναι μια συζήτηση που αφορά όλη την κοινωνία και θα πρέπει να υπάρχει βήμα συμμετοχή σε όλο τον αλευτικό τομέα. Επειδή έχει περάσει η ώρα, θα ήθελα να σταθώ σε κάποια μέτρα τα οποία έχουμε συμπεριλάβει στο έγγραφο στο οποίο αναφέρθηκα και τα οποία αναφέρθηκαν εν μέρη από τον συνάδελφο, τον γερουσιαστή ε, Τόρες, ο οποίος γνωρίζει καλά το λευτικό ζήτημα, διότι είναι και δήμαρχος της Σάντα Οχένια Ρεμπέιρα, μια πολύ σημαντική περιοχή στην Καρθία Δερόσα. Αυτά τα μέτρα, όπως υπενθύμηση και θα τα επαναλάβω εγώ, είναι το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτική πολιτικής θα πρέπει να έχει τρεις βασικές πτυχέ, τις κοινωνικές, τις οικονομικές και τις οικολογικέ πτυχέ. χωρίς όμως να δοθεί προβάδισμα σε καμία εκ των τριών ει βάρο των υπολείπων. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα διαφοροποιημένο καθεστώς για να προστατεύσουμε τις ε, παράκτιες ε, αλλιές, τον παράκτιο στόλο μικρής κλίμακας. Πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό το στόλο μικρής κλίμακας και θα το ήθελα να το επαναλάβω και εγώ εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έναν ορισμό. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε στόλος μικρής ε, κλίμακας. Επομένως, αυτός ο στόλος μικρής κλίμακας ε, θα πρέπει να προστατευθεί λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε αυτό στο οποίο αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι, τον κοινωνικό ιστό και ε, κάτι το οποίο αποτελεί παράδοση για πάρα πολλούς λαούς. Η σχετική σταθερότητα αναφέρθηκε επίσης. Εγώ θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στα ε, με τα βάσιμα δικαιώματα και για τον ε, ε, στόλο μεγάλης κλίμακας και επίσης ε, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να γίνει όχι μόνο διόρθωση στις αρχικές τιμές και στις τιμές οι οποίες καταβάλει ο καταναλωτές. Να σας υπενθυμίσω εδώ πόσο μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε. Αλλά επίσης θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε δυνατότητες για την βιώσιμη αλληλεία των κοινοτικών σκαφών μέσω των περιφερειακών οργανώσεων οργανώσεων Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γκαρσία Ντίεθ. Στη συνέχεια από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο κύριος Χάπτον από τη Σκοτία. Κύριε Χάπτον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως το είπατε και εσείς, Εκπροσωπώ εδώ το αλλιευτικό έθνος της Σκοτίας που αντιπροσωπεύει περίπου 70% των αλλιευτικών συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα σκοτικά χωρικά ύδατα περιέχουν, ε, είναι το 20% των ενωσιακών υδάτων και ίσως να σας εκπλήξει το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε εκπροσωπηθεί Στο Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια υπάρχουν πολλές τοπικές εκλογές, αλλά δυστυχώς από την εμπειρία μου και την εμπειρία των πρωτοκατόχων μου ξέρω ότι δεν είναι τίποτα καινούριο η διαπίστωση ότι οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δεν δίνουν προτεραιότητα στην εκπροσώπηση των αλλιέων ούτε στα συμφέροντά τους. Εδώ ακούσαμε σχεδόν τον καθένα να λέει ότι η περιφερειακή διαχείριση είναι καλή ιδέα με διαφορετικές απόψεις βέβαια ως προς το τι ακριβώς εννοεί αυτό. Ακούσαμε πολλά για το δικαίωμα μεταβίβασης δικαιωμάτων, ε, και τα λοιπά ποσοστώσεων και εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα δικαιώματα όπως τα προτείνει η Κομισιόν και η Επίτροπος μας διαβεβαιώνει ότι θα τύχει το σύστημα αυτό προστασίας εθνικός. Εμείς φοβούμαστε ότι εάν σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμοστούν αυτά τα μεταφερόμενα δικαιώματα σε πολύ λίγο χρόνο θα ακουστεί αφού έχουμε ενιαία αγορά πρέπει να είναι και διεθνώς μεταφέρσιμα τα δικαιώματα αυτά η Δανία ακούστηκε ως υπόδειγμα για τα δικαιώματα αυτά και τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα αλλά το σύστημα αυτό δεν ήταν ενωσιακό ήταν ενδοδανεζικό σύστημα τώρα για τις μικρής κλίμακας αλληλεία πρέπει φυσικά να προστατευθούν οι μικροί στόλοι και οι αλλιευτικές κοινότητες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν σε ενωσιακό επίπεδο να οριστούν, να οριστεί τι ακριβώς είναι μικρής κλίμακας στόλος και κοινότητα. Στην Κύπρο ας πούμε μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό ο μικρός στόλος από ό,τι στη Σκοτία μια μικρή κοινότητα με χαμηλό πληθυσμό στη Σκοτία μπορεί να στηρίζεται από ένα μικρό αριθμό σχετικά μεγάλων πλοίων, μεγαλύτερων από ό,τι στην Κύπρο ή στη Μάλτα. Ας αφήσουμε λοιπόν τα αλλιευτικά έθνη από μόνα τους να ορίσουν τι πρέπει να προστατευτεί. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε να υπάρξει ζωνική διαχείριση και να αφήσουμε τα αλλιευτικά έθνη που έχουν αλλιευτικά δικαιώματα εκείνα να καθορίσουν τι μέτρα θέλουν και θεωρούν ότι πρέπει να ληφθούν διατήρησης και συντήρησης. Διότι εκείνα έχουν το μεγαλύτερο συμφέρον από τα προγράμματα αυτά και η αξιότιμη πρόεδρος κυρία Φράγκα στη συζήτηση που έγινε με τον κύριο Καντέκ διαπίστωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να πετύχει μια κοινή πολιτική. Πολύ το σωστό είναι αυτό. Το είδαμε και στη Σκοτία, το αποδείχτηκε ότι είναι πολύ δύσκολο. Καλό θα ήταν λοιπόν να δοθούν πραγματικές δικαιοδοσίες και εξουσίες στις ίδιους τους ενδιαφερόμενους που έχουν τα καλύτερα δυνατά κίνητρα για να εφαρμόσουν μια επιτυχή πολιτική διατήρησης του μέλλοντος τους εγγύησης του μέλλοντος Και αυτό είναι μια επιλογή. Στη συνέχεια, από πλευράς Ισπανίας, ο Ντόν Βινθιέντε Γιάννος. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ παρεμβαίνω εξ ονόματος της Γερουσίας της Ισπανίας, ανήκω στην Επιτροπή Γεωργίας και Αλίας της Γερουσίας και θα ήθελα να τονίσω την κοινωνική πτυχή που ε, περιέχει η πράσινη βίβλο σε σχέση με τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτικής πολιτική. Σε σχέση με άλλα θέματα που αναφέρονται στην πράσινη βίβλο θα πρέπει να τονίσουμε την κοινωνική πτυχή τη κοινή αλληλευτική πολιτική και την ανάγκη αναζήτηση κάποιων δυνατοτήτων, ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και την ε, συμμετοχή των νέων στον τομέα αυτό. Η ανάγκη διατήρηση σταθερών ε, προποθέσεων για τα πληρώματα ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της ελεκτικής πολιτικής. Όσον αφορά τη μετατοκαλλιέργεια, η συνεχής ε, ζήτηση για τέτοια προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα, πάνω από τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των θαλασσών, επιτρέπει να προβλέψουμε ότι η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να μετατραπεί στην, ε, σε απάντηση σε αυτή την υπάρχουσα ζήτηση. Υπό την έννοια αυτή η ισπανική ε, ε, κυβέρνηση είναι υπέρ του προγραμματισμού μιας βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας συμβατής με το περιβάλλον που να εγγυάται στους καταναλωτές ορισμένα προϊόντα υψηλού επίπεδου υγιή και ασφαλή. Η Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα τη στρατηγική τη σε αυτό το τομέα μέσω μια ανακοίνωση που απευθύνεται προ το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον τη εδατοκαλλιέργεια που έχει τρεις ε, άξονες ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της ε, εικόνας της διακυβέρνησης. Για να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη της δατοκαλλιέργειας μαζί με τους άλλους ε, κλάδους της αλίας και να εγγυηθεί ο ρόλος που θα πρέπει να διαρματίσει στο μέλλον η δατοκαλλιέργεια θα πρέπει να συμπεριληφθεί πλήρως στο μέλλον της κοινή τη κοινή ε, πολιτικής. Γιατί είναι σημαντικό πυλώνας τη. Υπό την είναι ευθύνη αναγκαίο να αναπτυχθούν τα αναγκαία μέτρα ούτω ώστε η δατοκαλλιέργεια να συμπεριληφθεί στον ΠΟΕ με το ίδιο επίπεδο expectation ε, όπως και η λυπή αλία. Ε, είμαστε υπέρ της υποστήριξης μέσω κονισιών αυτής της πρωτοβουλίας. Για να κλείσω θα ήθελα να αφερθώ στα θέματα σχετικά με τον αληφτικό στόλο και θα ήθελα να μνημενεύσω την παράκτια αλία μικρής κλίμακας που θεωρούμε ότι είναι αναπόσπαστη διάσταση της επιβίωσης ε, του αλληλευτικού κλάδου. Και εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, τα ζητήματα ενίσχυσης των παράκτιων ε, ζωνών, η συμπερίληψη των νέων στον κλάδο και η κατάλληλη κατάρτισή τους. Επίσης, η διατήρηση ορισμένων κατάλληλων προϋποθέσεων για την επαγγελματική άσκηση της παράκτειας αλίας μικρής κλίμακας με παράλληλες εγγύησεις ασφαλείας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιάννου. Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο η κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ε, προσκεκλημένους μας. Έχουμε κάνει πολλές ε, συνεδριάσεις τέτοιου τύπου και αυτό δείχνει ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει στη διαδικασία συναπόφασης. Και οι προσκεκλημένοι μας βλέπουν πόσο σοβαρά παίρνουμε αυτό το θέμα. Εμένα με εντυπωσίασε ο συνάδελφος από τη Σουηδία, ο οποίος είπε ότι μόνο μέσω κοινωνιολογικής ε, δράσης ε, καθίσταται δυνατή η κοινωνιοοικονομική οικονομικη δράση. Νομίζω ότι αυτή είναι η σημαντικότερη φράση που διατυπώθηκε εδώ. Μόνο με την πρόθεση μιας βιώσιμης αλίας θα είναι δυνατό να υπερασπιστούμε αυτό το δημόσιο αγαθό περί το οποίο μιλούμε, ούτως ώστε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να μπορούν να συνεχίσουν να τρώνε ψάρια. Γιατί μιλούμε για ένα δραματικό αριθμό που αναφέρει το ΒΒΕΦ, πάνω από 80% υπεραλίευση. Και ε, συνεπώς το βασικό μας μέλημα είναι η οργάνωση της βιωσιμότητας και η διατήρηση της βιωσιμότητας γιατί τελικά μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν ε, θέσεις εργασίας και να επιβιώσει ο πολιτισμός της παράκτιας αλίας. Ε, έγινε μνήα στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Βλέπουμε στην τηλεόραση τι γίνεται όταν υπάρχει έκρηξη μιας ε, πλατφόρμας εξόριξης ε, πετρελαίου. Για μένα η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική δεν θα πρέπει να ασχολείται μόνο με ζητήματα μεταφορών, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τη χάραξη τη πολιτική αλλία. Τώρα, όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, αυτό έχει, ε, τέθηκε κατά επανάληψη. Μιλούμε πάνω από 10 χρόνια για θέματα αυτά, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι παρόλα αυτά ότι στην Ευρώπη ε, το θέμα αυτό βρίσκεται στα σπάργανα ακόμα. Χρειαζόμαστε έναν ε, δεσμευτικό κανονισμό που να συνδέεται επίση και με την προστασία των ε, ζώων. Θα πρέπει ε, επίσης να περιμνήσουμε να μην ε, ζημιωθεί και ο τουρισμός. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο τέθηκε εδώ κατά επανάληψη, το ζήτημα της έρευνας. Εδώ απομένουν πολλά να γίνουν. Θα πρέπει να κατασκευάσουμε κάποιες, κάποια λεφτικά μέσα τα οποία να είναι συμβατά με τις ε, περιβαλλοντικές προδιαγραφές και για να γίνει αυτό χρειάζονται χρήματα. Επίσης η βιωσιμότητα που θέλουμε να αναπτύξουμε ε, προϋποθέτει ε, αποτελεσματικούς ελέγχους. Ελέγχουμε αποτελεσματικά. Όχι. Με τους ελεγκτές που έχουμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο ο αριθμός είναι εξαιρετικά περιορισμένος, δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί απολυσματικό έλεγχο. Γι' αυτό θα πρέπει οι Υπουργοί Οικονομία να σκεφτούν κατά πόσο δεν θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα κονδύλια στου ελέγχου. Ω, λέει ο μιλήτρια, ξεπέρασα το χρόνο μου, αλλά θα τα βρείτε αυτά. Ε, στην ε, έκθεσή μας. Η συνάδελφος κυρία Περέιρα ήταν ε, σκιώδης ε, εισηγήτρια και πραγματικά μπόρεσε να συμπεριλάβει τα, την άποψη της σοσιαλιστικής ομάδας. Ο κύριος Στίξλιν από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφός μου Λάρσον έλαβε το λόγο προηγουμένως και την, τον συνεχάρει η Γερμανίδα συνάδελφος. Για να δω αν θα με συγχάρει και εμένα. Λοιπόν, η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά και μένα με ανησυχούν ορισμένες ιδέες. Έχω την εντύπωση ότι εδώ μοιράζουμε πόρους που δεν τους διαθέτουμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι, ότι λέγω 8 στα 10 Ήδη που αλλιεύονται στα ενωσιακά ύδατα, αλλιεύονται στα ενωσιακά ύδατα και με αυτό οι επιχορηγήσεις που δίνονται, δίνονται από τον φορολογούμενο και τη φορολογούμενη. Η Επίτροπος λέει ότι δεν θέλει πια να πληρώνει η Ένωση τον παροπλισμό των στόλων αλλά ελπίζω να σταματήσει και η αλίευση σε ξένα χωρικά ύδατα και η κατασπατάληση των καυσίμων. Γιατί βέβαια κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει ούτε όμως και να επιβάλλει τη χρησιμοποίηση ακαταλήλων μηχανών και την εφαρμογή μιας μη βιώσιμης αλληλείας. Αυτά είναι πράγματα που είναι απαράδεκτα πρέπει να επιμείνουμε για τη διατήρηση των αλλιευτικών πόρων. Σήμερα η πολιτική βασίζεται πια σε τρεις πυλώνες, πολιτικό, κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ούτε έναν από τους τρεις. Μέχρι τώρα η κατάσταση δεν χαρακτηριζόταν από ισορροπία και γι' αυτό φτάσαμε στην καταστροφή επαναλαμβάνω, οικονομία, περιβάλλον και κοινωνική πτυχή. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κανέναν από τους τρεις παράγοντες. Το ίδιο ισχύει και για τις ποσοστώσεις. Εφόσον λέμε ότι τα ψάρια είναι δημόσιος πόρος, τότε πώς τα πουλάμε. Πώς τα πουλάμε. Μπορούμε να τα αλλιεύουμε αλλά όχι να τα πουλάμε. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιφάσεις αλλά και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που ακούστηκαν. Και η υδατοκαλλιέργεια είναι και αυτή κάτι το ενδιαφέρον, αλλά τίθεται άλλο ερώτημα. Με τι θα ταΐζουμε τα ψάρια στις υδατοκαλλιέργειες, με άλλα ψάρια πρέπει να γίνει έρευνα και να επιδειχθεί μεγάλη φρόνηση ως προς το σε τι θα επενδύσουμε, τι θα πληρώσουμε δηλαδή. Έγινε λόγος για απαγόρευση των απορρίψεων, σημαντικό μεν θέμα, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι η βιωσιμότητα, η οικολογική βιωσιμότητα της αλληλείας. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όμως αν πετύχουμε τη βιωσιμότητα θα τα έχουμε λύσει όλα. Η συμβουλή που σας δίνω λοιπόν είναι να τα ρίξουμε, να ρίξουμε όλο το βάρος στη βιωσιμότητα. Ο κύριος Κούν, Γερμανός βουλευτής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι, ένα πολύ σημαντικό, είναι πολύ αυτό το φόρουμ που έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με του περιφερειακού πολιτικού, γιατί είναι αναγκαίο να γίνουν εδώ ορισμένε διευκρινήσει. Και θα ήθελα να απαντήσω στην επιχειρηματολογία των πρασίνων που λένε ότι δεν συζητούμε ή δεν κρίνουμε ε, στη βάση επιστημονικών δεδομένων και ότι είναι μόνο πολιτικές απόψεις. Όχι. Δεύτερον, λέγεται ότι τα αποθέματα υπεραλλιεύονται, αλλά εμείς ως πλούσια Ευρώπη επιτρέπουμε στον αυτού μας μια υπερβολική προστασία ειδών Ιδιαιτέρως ε, στα ύδατα της ε, Βόρειας Θάλασσας, κάτι που δεν έχει τον όμοιό του πουθενά στον πλανήτη. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Είμαστε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας με 5 εκατομμύρια κατοίκους σε ψάρια ε, και καταναλώνουμε 4 εκατομμύρια τόνους ανά έτος. Οι προδιαφθέσεις που έχουμε είναι ιδιαίτερα υψηλές. Και βεβαίως αυτό είναι ορθό γιατί θα πρέπει να προσέχουμε τις αγωγές. Αλλά από την άλλη πλευρά μίλησα για μια υπερβολική προστασία των ειδών. Και θα πρέπει να δούμε. Και υπάρχουν εδώ οι συνάδελφοι από τις χώρες της Βαλτικής, ε, της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Ε, τι κατανάλωση ψαριών έχουν εκείνοι και τι απαγορεύσεις υπάρχουν ή ε, τι είπε ο συνάδελφο από τη Σλοβακία, ποιε είναι οι ζημιέ που κάνει Κομοράνη, παρόλο που δεν είναι πια αποελούμενο είδο. Και ο συνάδελφο από την ε, Σουηδία επίση ε, θα πρέπει να συμφωνήσει όταν μιλούμε για το μέγεθο και του πληθυσμού από Και είναι 100.000, αν όχι ένα εκατομμύριο τόνοι ανά έτος, που για να θρέψουμε ε, αυτά τα είδη τα οποία δεν ε, απειλούνται πλέον. Πρόκειται για υπερβολική προστασία ειδών. Ε, νομίζω ότι πρόκειται για τεράστιες αντιφάσεις εδώ. και όσα, όσον αφορά την, την γερμανική αλληλευτική πολιτική αναφέρθηκε σχετικά η κυρία Ρούμφα. Και τώρα θα, ήθελα να κατεβάσω τους τόνους και να πω ότι η Ευρώπη είναι μια υπέροχη ήπειρος που έχει χιλιάδες ε, χιλιόμετρων ακτογραμμής και ο ποτηρισμός είναι ιδιαίτερο σημαντικός. Και η διασύνδεση μεταξύ ε, παράκτιας αλίας μικρής κλίμακας και ιστορικής παράδοσης στην αλία με τον τουρισμό είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό θέμα και αυτό το τομέα θα πρέπει να τον στηρίξουμε και να τον προωθήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Κούν. Και τώρα ο τελευταίος ε, αγορητής από πλευράς προσκεκλημένων μας, ο κύριος Τροτσικόσκι από την Πολωνία. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε πολλές ε, σημαντικές παρατηρήσεις στα πλαίσια της σημερινής συζήτησης. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα έχουμε ήδη ακούσει σήμερα στα θέματα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Μία σημαντική παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διαχείριση, κατάλληλη διακυβέρνηση και θα πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία. Γεγονός που πιστεύω ότι σημαίνει ότι η περιφερειοποίηση θα πρέπει να γίνει επί τη βάση κατάλληλης επιστημονικής γνωμοδότησης για να λαμβάνουμε και τις κατάλληλες αποφάσεις. και θα πρέπει να δίνονται και ε, δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να επηρεάζουν αποφάσεις που τους αφορούν. Μπορούμε να κάνουμε πολλά αν συνεργαστούμε. θα υπάρχουν αποφάσεις λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας και τα τοπικά και περιφερειακά επίπεδα διακυβέρνησης έχουν συγκεκριμένα τοπικά ε, στάνταρ τα οποία μπορεί να έχουν και κάποιες θετικές επιπτώσεις. Νομίζω ότι αυτά που ακούσαμε σήμερα ε, θα εισακουστούν και εκτός εθούσης και νομίζω ότι αυτή είναι μια θετική και επικοδομητική προσέγγιση. Άκουσα πολλούς εδώ στην αίθουσα να μιλούν για την ανάγκη να φροντίσουμε τις, την μικρή κλίμακα παράκτη αλία και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη φροντίδα τους. Οι αλληλείς βρίσκονται στη ρίζα του κλάδου, αν θέλετε, και θα πρέπει να μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε, γιατί αλλιώς οι μεγάλες επιχειρήσεις θα καταστρέψουν κάθε δυνατότητα μικρής κλίμακας αλία στις παράκτητες περιοχές. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή άγουσα και θα πρέπει να αποφύγουμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, βλέποντα τι πρακτικές ακολουθούμε. Και τώρα, κυρία Παρτήρο, τώρα θα μιλήσω εγώ ως Ευρωβουλευτής, όχι ως Πρόεδρος. Ναι. θα ήθελα να πω τα εξή. Θα ξεκινήσω από μία φράση της κυρίας Πατράο Νομίζω ότι η μεταρρύθμιση αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερική πολιτικής αν θέλουμε η Αλία να συνεχίσει να είναι μια δραστηριότητα που θα διατηρηθεί και στο μέλλον. Τα προβλήματα της αλληλείας, ε, νομίζω ότι τα αναγνωρίζουν όλα, είναι η υπεραλίευση και οι ε, υπερβολικές ε, δυνατότητες. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του υπολείπου κόσμου. Και νομίζω ότι σωστά το επισήμανε και η ΦΑΟ αυτό. Και αυτό ήταν και η μεγάλη αποτυχία του συστήματος διαχείρισής μας. Όλοι αναγνωρίζουν ότι απέτυχε το προηγούμενο σύστημα και με εκπλήσει το γεγονό ότι κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν να το διατηρούν. Χρειαζόμαστε πιο ευέλικτα μοντέλα και αυτό το είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χρειαζόμαστε και πιο ευέλικτα μοντέλα τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν δύο πτυχές πολύ σημαντικές κατά με. Να είναι εύκολα στη διαχείρισή τους, γι' αυτό ακριβώς και εμείς δεν είμαστε υπέρ του συστήματος ε, ελέγχου αναλυτική προσπάθεια και δεύτερον, για τα συστήματα διαχείρισης, όπως αυτά τα οποία ανέφερε η Επίτροπος, ε, δικαιωμάτων ε, μεταφοράς μεταβιβασμένων δικαιωμάτων όπως αυτά που είπε η Επίτροπος και είναι αυτά τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε όλο και πιο ανταγωνιστικοί σε ε, μια όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Οι στόλοι οι οποίοι θα πρέπει να έχουν και μια βιομηχανική δομή και θα είναι πιο ανταγωνιστικοί είναι οι στόλοι οι οποίοι μπορούν να παραμείνουν και είναι και αυτοχρηματοδοτούμενοι. Δεν θα εξαρτώμεθα από τη δημόσια χρηματοδότηση, διότι η δημόσια χρηματοδότηση, όπω πολύ σωστά είπε η Επίτροπο, θα σταματήσει για πολλού λόγου που μα είπε η αλλά και για λόγου που έχουν να κάνουν και με την προσωπική μας συμμετοχή στον ΠΟΕ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμβεί και αυτοί που είναι υπέρ του, διαχειρι... του συστήματος διαχείρισης βασίζονται σε ένα μοντέλο δημόσιας χρηματοδότησης που είτε το θέλουμε είτε όχι θα σταματήσει. Η κάνουλα θα κλείσει και θα γίνει για πολύ συγκεκριμένου λόγους και για πολύ συγκεκριμένου τόλους που δεν μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε δυνατότητες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ε, στους στόλους που μπορούν, ε, συστήματα Όπω το ITR, το οποίο συστήνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από το ΦΑΟ και από την ΩΣΑ, διότι είναι μοντέλα τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικά από οικονομική πλευρά και μειώνουν και το πρόβλημα τη υπεραλίευση, που είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε και δεν έχουμε καταφέρει να το επιλύσουμε ακόμα και μέσω τη δημόσια χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ελαστικοί, να δείχνουμε περισσότερη κατανόηση και να κατανοήσουμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα διαχείριση και να το προσαρμόσουμε και στου τόλου αλλά και και στα διάφορα είδη αλίας. Και από εκεί και πέρα και στην ε, χρηματοδότηση που θα πρέπει να αυτοχρηματοδοτείται και θα, θα περιορίζει τις επιδοτήσεις. Θα σταματήσω εδώ για να μην ε, μιλήσω περισσότερο από τους υπολείπους και θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 5 λεπτά και μετά στην κυρία Πατράο Νέβες και μετά θα κλείσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Πένιας έχει το λόγο και στη συνέχεια θα τελειώσει κυρία Πατράου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέλο πάντων, εγώ θα ολοκληρώσω, αλλά τέλο πάντων, πέντε λεπτά ο καθένα. Και μετά θα μου δώσετε τρία λεπτάκια για να ολοκληρώσω τη συζήτηση. Κύριε Πένια, ω καλό υπάλληλο μπορείτε κάλλιστα να μα κάνετε μία σύνοψη και νομίζω ότι θα μπορέσετε να απαντήσετε και στην πλειονότητα των ερωτήσεων σε πέντε λεπτάκια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω και σε πολλέ ερωτήσει αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα ήθελα ήταν να επαναλάβω τα λεγόμενα τη Επιτρόπου και να πω ότι είναι απαραίτητο να διαθέτουμε ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έχει ο λευτικός τομέας για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα ισχύει για τη διαχείριση της αλίας μόνο για το 2013, αλλά θα πρέπει να είναι και το κατάλληλο ώστε να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές, να αντιμετωπίσουμε τις κατάλληλες προκλήσεις και τα προβλήματα τα οποία θα έχει η ευρωπαϊκή ε, αλληλεία μέχρι το 2020. Σε αυτό αναφερόμαστε. Και εδώ θα πρέπει να πω κυρία Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε μια πλήρη διαδικασία περισυλλογής. Ε, νομίζω ότι τα είπε και η κυρία Δαμανάκη πολύ σωστά. Δεν έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες παγιωμένες θέσεις. Ε, μόνο αυτά τα οποία σας είπε η ίδια είναι σταθερά. Όσον αφορά στα περισσότερα θέματα, είμαστε σε μια διαδικασία που πραγματικά μας ενδιαφέρει να ακούσουμε οποιαδήποτε ιδέα μπορείτε να μας προσφέρετε. Έχουμε σημειώσει πολλές πολύ καλές ιδέες ε, στη διάρκεια αυτής της συζήτηση και όλα αυτά θα τα αναλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ε, μέγιστη δυνατή προσοχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πατράων Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτησα το λόγο μου υπό την ιδιότητά μου ως ε, Πορτογαλίδας ε, υπηκόου ορισμένοι συνάδελφοι μου έδωσαν κάποια εξουσία ως συγκήτρια. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή τις ευκαιρίες να πω ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ζώνη αλίευσης ε, στην ε, Ευρώπη. Δεν είναι εντυπωσιακό λοιπόν το γεγονός ότι η μείωση του στόλου ήταν ιδιαίτερο οξύ πρόβλημα στη χώρα μου αλλά η πρόεδρος μου έδωσε το λόγο σε αυτό το τελικό στάδιο της συζήτησης ως εισηγήτρια. Και θα έλεγα ότι βρήκα αυτό το απόγευμα, αυτή την απογευματινή συνεδρίαση ιδιαίτερως ε, ενδιαφέρουσα και αντανακλά την πλατιά συνένεση που είχα ήδη διαπιστώσει προηγουμένως. Γιατί όλοι έχουμε συνείδηση ότι είναι ένα ε, ιδιαίτερο σημαντικό έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ο δρόμος θα είναι τραχής, θα πληρώσουμε ένα ψηλό τίμημα και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλο μας το θάρρος για να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Ωστόσο θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα το οποίο ανέκυψε με αρκετά προφανή τρόπο και πρόκειται για τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα τα ITR, ε ένα θέμα επίμαχο. Ακόμα και το θέμα αυτό θα μπορούσε να λυθεί καλύτερα εάν αφιερώμε μεγαλύτερη ε, προσπάθεια στο ζήτημα της περιφερειοποίησης. Αν είχαμε ένα ισχύον ε, μοντέλο περιφερειοποίησης, το οποίο είναι αρκετά περιεκτικό, θα μπορούσε να λυθεί. Γιατί θα μπορούσαν να δοθούν πιο ευνοϊκέ λύσει, για παράδειγμα προ τα διαχειριστικά μοντέλα. Ναι, χρειαζόμαστε κάποια περιθώρια ευελιξία. Δεν μπορεί να ισχύουν όλα τα μοντέλα για όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Αλλά ποιο θα έχει τον τελευταίο λόγο όταν το ζητούμενο είναι η λήψη αποφάσεων. Εάν έχουμε μια αποτελεσματική περιφερειοποίηση, τότε οι αποφάσεις αυτές μπορούν να γίνουν με έναν αποκεντρωμένο τρόπο. Και αυτό ισχύει επίση για την ε, διάκριση μεταξύ βιομηχανικού και στόλου και στόλου